Okay, colleagues, give you a lot of leeway for first committee since, um, since, since Christmas Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι η πρώτη μας συνεδρίαση μετά τις ε, χειμερινές κοπές, αν και είχαμε άλλες ευκαιρίες να συναντηθούμε. Σας εύχομαι πάντως καλή χρονιά. Ελπίζω να είναι και επικοδομητική χρονιά το 2015, Ευρωπαϊκό έτος της ανάπτυξης όπως γνωρίζετε, το οποίο με επιτυχία το οποίο με επιτυχία και η έναρξη στη Ρήγα πριν από λίγες μέρες. Θα μας το πει ασφαλώς και η εκπρόσωπος της Προεδρίας. Το έχουμε και στην ημερήσια διάταξη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την κήρυξη της έναρξης του Ευρωπαϊκού Έτσου Ανάπτυξη. Έχουμε και άλλα θέματα όμως χρηματοδότησης με τον Ερικ Σόλχαϊμ. Πολύ σημαντικό μιλητή, τον οποίο συνάντησα και στη Ρήγα και έχει να μας δώσει πολλές ιδέες για πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη. Πριν περάσω στο, όμως στον κύριο Σολχάιν που θα μας μιλήσει για το πρώτο σημαντικό θέμα της μέτρησης διάταξης, θα περάσω στο σχέδιο, το υπαριθμόν 1, έγκριση λοιπόν της μέτρησης διατάξεως, παρατηρήσεις δεν υπάρχουν, δεύτερον έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, έχετε τα πρακτικά της 10-11 Νοεμβρίου, 17 Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου στα πρακτικά σας. Εάν έχετε παρατηρήσεις παρακαλούμε να ενημερώσετε τη γραμματεία έως το τέλος συνεδριάσεως. Αν μέχρι τότε δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις παρατηρήσεις θεωρείτε ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Στο σημείο 3. Έχουμε την έκρηση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών τη 11η Νοεμβρίου και τη 10η Δεκεμβρίου 2014. Και πάλι, αν έχετε κάποιε παρατηρήσει, παρακαλώ να με ενημερώσετε. Ή θα άλλω θεωρούνται εγκεκριμένα. Ανακοινώσει δεν έχω. Θα δώσω όμω το λόγο στο 5 τη σημερινή διάταξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα παρακαλέσω τον Πίτερ Κρέικ Μακουέι να μα πει αν έχει κάτι εκ μέρου τη Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ στόμα να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα και άλλωστε το συζήτησε και το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Για το δικό μα πεδίο έχουμε ένα κύριο ζήτημα που καταγράφει το επίσημο πρόγραμμα εργασιών τη Επιτροπή. Θα ήθελα να σα το εκθέσω. Για τα υπόλοιπα σημεία δηλαδή τα οποία δεν περιλαμβάνουν το επίσημο πρόγραμμα εργασίας θα επανέλθω σε μεταγενέστερη συνεδρίαση μάλλον τον επόμενο μήνα. Από το πρόγραμμα εργασίας λοιπόν στο πεδίο της ανάπτυξης έχουμε την ανακοίνωση παγκόσμια εταιρική σχέση για την εκρίζωση της φτώχειας και την παγκόσμια ανάπτυξη μετά το 2017. Ξέρετε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών έχει υποβάλει έχει εκδώσει μάλλον μία συνθετική έκθεση και προχωρούμε προς τη σύνοδο του Σεπτεμβρίου με την προετοιμασία αυτής της ε, εκθέσεως. Έτσι λοιπόν από, για την περίοδο μετά το 2015 έχουμε μπροστά μας να ορίσουμε και να επιτελέσουμε βιώσιμους πόρους, ε, πόρου, πόρους και στόχους, το πλαίσιο και σχετικές διαδικασίες που είναι εν εξελίξη όπως αυτή που αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Η διάσκεψη του Ιουλίου στην Αντισαμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη χρηματοδότηση και τους τρόπους υλοποίησης της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης. Το Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2014 υιοθέτησε ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση παγκόσμιας εταιρικής σχέσης και να υιοθετήσει μια ενιαία συνεκτική ε, στεναρή θέση ενώπιση των διαπραγματεύσεων. Μετά λοιπόν ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Γενικών Υποθέσεων που επίσης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια συγκεκριμένη ε, στόχευση ενώπιση της παγκόσμια αυτής της εταιρικής σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε την ανακοίνωση με τις θέσεις μας, με τα κύρια σημεία, με το ρόλο που βλέπουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε για τους ε, βιώσιμους στόχους, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης από το 2015, περιβάλλον σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τομείς πολιτικής όπως ανάπτυξη δυνατοτήτων, έρευνα, επιστήμη, εμπόριο, επενδύσεις και δημόσιες, χρηματοδότηση ιδιωτική και δημόσια αλλά και διεθνής, αποτελεσματική αναπτυξιακή βοήθεια και δεσμεύσεις ε, όσο και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσμονές σε σχέση με την δράση των άλλων. Έχουμε επίσης ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης και ενώ γνωρίζουμε τι περιμένουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο θα ορίσουν η ανακοίνωση και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Πολύ σύντομα λοιπόν θα δημοσιευθεί η ανακοίνωση με στόχο να προσδιορίσει θεμέλια της ευρωπαϊκής στάσης και της πορείας ενώψη της Αντισαμπέμπα. Θα επανέλθουμε στις αρμόδιες αρχές του Κοινοβουλίου και θα συζητήσουμε περαιτέρω τα θέματα αυτά μαζί σας όταν είναι έτοιμη ανακοίνωση. Το πρόγραμμα εργασίας Επιτροπής, όπως σας είπα, είναι διαρθρωμένο με βάση τις 10 πολιτικές προτεραιότητες του Πρόεδρου της Επιτροπής Πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει και σε άλλες πολιτικές προτεραιότητες που έχουν να κάνουν και με την ενέργεια και με τη μετανάστευση στο θέμα της ανάπτυξης και άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί και τώρα μην αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας θα προκύψουν σύν το χρόνο και αυτά μπορεί να, να παρουσιαστούν στα άλλα θεσμικά όργανα σε μεταγενέστερο στάδιο. Ευχαριστώ. Και τι εννοείται σύντομα, λέει η κυρία Μακέβεν. Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο θα δούμε την ανακοίνωση. Ξέρω ότι θέλουν χρονοδιάγραμμα για τη δουλειά σου, συνάδελφοι. Πότε προβλέπετε να συνεδριάσει ο Συλλογικό Όργανο η Επιτροπή. Αναμένεται μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου να υιοθετηθεί η ανακοίνωση. Πάντως όχι πριν από τις αρχές Φεβρουαρίου. Ο κύριος Γκέρενς έχει μια ερώτηση πολύ Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Κατά τη διάρκεια του 2015 σκοπεύει να υποβάλει καινούριε προτάσεις ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για τη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα. Τρεις χώρες που πλήττονται από τον, την πανδημία του έμπολα. Με 10% της ανάπτυξής τους κάτω από το αναμενόμενο εξαιτίας του έμπολα. Ε, θα εξετάσουμε τη δυνα... τις οικονομικές δυνατότητες των χωρών αυτών, τη δυνατότητα απορρόφησης της βοήθειας και πότε να περιμένουμε προτάσεις αν σκοπεύει η Κομισιόν να εξετάσει το πρόβλημα. Δεν γνωρίζω την απάντηση. Θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Περνάμε στο σημείο 6. Ε, μας είπε η Κομισιόν ότι ετοιμάζει για την Αντισαμπέμπα ε, και για τον Σεπτέμβριο ε, ετοιμάζεται μάλλον για την Αντισαμπέμπα και για τον Σεπτέμβριο έχουμε τον Έρικ Σόλχαϊτ μαζί μας είναι πρόεδρος της Επιτροπής DAC δηλαδή Αμυσιακής Βοήθειας του ΟΣΑ η... την κυρία Τον κύριο Σολχάιμ, ε, τον ε, είχα δει στην ε, ε Ρίγα ε, και χαίρομαι που θα τον ξανά έχουμε εδώ μαζί μας. Η Επιτροπή μας θα είναι πολύ σημαντική τις επόμενους μήνες γιατί θα πρέπει να απαντήσει το ανακοινωθέν της Κομισιόν οπότε θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε την άποψη του ΩΣΑ. Να μπορείτε να μας πείτε τι κάνει όσα και να συνεισφέρετε έτσι και στις δικές μας εργασίες. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας με τον κύριο Ντέβα και με άλλους συναδέλφους ξεκινήστε να συνεργάζεστε με την κοινωνική κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, ε, με τον κύριο Ντεβακή, για αυτό το θέμα είχαμε συνεργαστεί. Ε, στην Σρι Λάνκα έχει αρχίσει η ανοικοδόμηση της χώρας, ε, οικονομική ανοικοδόμηση με αύξηση του τουρισμού με την, και με προσπάθειες ειρήνευσης με την μειονότητα των Ταμίλ. Θα πρέπει να προσκληθούν στις Βρυξέλλες και σε όλες τις πρωτεύουσες ε, προκειμένου να τους βοηθήσουμε με επενδύσεις ε, έχουμε πολλά δύσκολα ε, πολλά εμπόδια που θα πρέπει να υπερπηδηθούν. Τώρα αυτό δεν έχει σχέση βέβαια με την δική μου παρουσίαση αλλά χρειάστηκε να σας το πω. Είναι όχι απλώ το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, αλλά το Έτος Ανάπτυξης το 2015. Έχουμε, ε, έχουμε το Σεπτέμβριο τη Νέα Υόρκη, τη διάσκεψη του Παρισιού για, το, για την κλιματική αλλαγή επίσης. Ε, όλα αυτά θα μας υπαγορεύσουν, θα μας υποχρεώσουν να πάρουμε αποφάσεις φέτος που θα περάσουν τα επόμενα χρόνια. Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, να θυμηθούμε ότι είμαστε πάρα πολύ πετυχημένοι στον τομέα της ανάπτυξης. Όταν βλέπουμε τηλεοράση, στην τηλεόραση εικόνες από το Ιράκ, από την Ουκρανία κλπ. Ε, κανείς νομίζει ότι κινούμαστε προς τον κρεμό. Όμως στην ανάπτυξη σημαίνει το αντίθετο ακριβώς. Έχουμε τρομακτική επιτυχία τα τελευταία δέκα χρόνια. Ε, έχουμε μειώσει την φτώχεια στο μισό. Ε, έχουμε μειώσει στο μισό τα, τον αριθμό των παιδιών που πεθαίνουν. Ε, όλα αυτά είναι τα θετικά της αντισυχιακής βοήθειας. Έχουμε εξασφαλίσει περισσότερο πλούτο, περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη ευημερία σε όλο τον πλανήτη από ό,τι ποτέ στην ιστορία μας. Είμαστε πετυχημένοι λοιπόν στην αναπτυξιακή βοήθεια και θα πρέπει να επιταχύνουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρουμε τι είναι αυτό που φέρνει ανάπτυξη και ξέρουμε τι είναι αυτό που μας κάνει να αποτυγχάνουμε. Πολύ παλιότερα, το δεκαετία του 60 70, δεν είχαμε αυτή τη γνώση. Ε, μόνο η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν πετύχει την ανάπτυξή του. Τώρα έχουμε σημαντικέ επιτυχίε σε όλο τον κόσμο, σε όλε τι πύρου. Ξέρουμε τι είναι αυτό που φέρνει ανάπτυξη. Πριν ε, επισέλθω στα οικονομικά τη ανάπτυξη, να σα υπενθυμίσω ότι το υπαριθμόν ένα θέμα είναι οι πολιτικοί, οι σωστές πολιτικές και όχι τα οικονομικά. Ε, οι σωστές πολιτικές μπορούν να μας σώσουν. Και τα όσα συνέβησαν στην Κίνα μετά το 1970 είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και επετεύχθη με την αλλαγή της κυβέρνησης, με την αλλαγή της πολιτικής. Αν δεν είχε γίνει αυτό, εκείνα θα βρισκόταν, θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Πηγαίνετε στην Κορέα, στο, στα σύνορα μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Εκεί θα δείτε τη διαφορά. Η Νότια Κορέα είναι 390 φορές πιο πλούσια κατά κεφαλήν από το 1950. Εκπληκτική επιτυχία. Την Βόρεια Κορέα από την άλλη μεριά έχουμε παιδιά που πεινούν ε, μια βάρβαρη δικτατορία και φτώχεια παντού εκτό από μερικού ελάχιστους πλούσιους. Ποια είναι η διαφορά? Δεν είναι η κουλτούρα, δεν είναι η θρησκεία, δεν είναι η ιστορία. Έχουν περισσότερες πρώτε ύλε στον Βορρά για να καταλάβετε. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν? Η Νότιος Κορέα πήρε τι ορθές πολιτικέ αποφάσει. Όχι όλε. Δεν ήταν όλε οι αποφάσει σωστέ. Αλλά σε μεγάλο βαθμό οι πολιτικέ του αποφάσεις ήταν σωστέ και στο βορρά ήταν λάθο. Αυτή ήταν η διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι η Νότιο Κορέα βοηθήθηκε πολύ από την Δύση κατά τη διάρκεια του πολέμου τη κορέα, αλλά ήξεραν πώ να τη χρησιμοποιήσουν αυτή τη βοήθεια. Μπορώ να δώσω και πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενό μου σήμερα να μπω στα οικονομικά της ανάπτυξης. Και τα οικονομικά όμως θα βοηθήσουν πραγματικά μόνο αν τεθεί το σωστό πολιτικό πλαίσιο. Έτσι, ναι, μπορούν να βοηθήσουν και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία, η Νότιος Αμερική, η Κορέα, η Κίνα, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Ινδονησία, όλες αυτές είναι τεράστιες επιτυχίες. Ε, η Ινδονησία έχει τριπλασιάσει το κατακεφαλήν ΑΕΠ της τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα. Έχουμε τρεις βασικές πηγές χρηματοδότησης. Βοήθεια, φορολογία και ιδιωτικές επενδύσεις. Και δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ αυτών των τριών. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίφαση Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη ιδιωτική επένδυση, καλύτερους και περισσότερους ε, φόρους, καλύτερη συλλογή και περισσότερους φόρους και βέβαια περισσότερη ε, δωρεάν βοήθεια. Ας ξεκινήσω από τη βοήθεια. Η, η κοινότητα, η κοινότητα σε όλο τον κόσμο μιλάει μια γλώσσα λίγο πεχειωμένη. τίθεται το θέμα του κατά πόσον η βοήθεια είναι το πιο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Ε, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά δεν είναι το βασικό εργαλείο. Ο ΣΑ θέλει να αναμορφώσει την αναπτυξιακή βοήθεια και το σύστημά της για να την προσαρμόσει στη σημερινή πραγματικότητα. Πρέπει να εστιάσουμε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Γιατί αυτές οι χώρες έχουν λιγότερες εναλλακτικές λύσεις, δεν μπορούν εύκολα να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, για παράδειγμα. Θα πρέπει να εστιαστούμε λοιπόν, να εστιάσουμε την ε, ε, ενθουσιακή μας βοήθεια κυρίως στην Αφρική, ε, αλλά και κάποιες άλλες, ε, κάποια άλλα σημεία του κόσμου όπως η IT για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε καλύτερα εργαλεία που να είναι προσαρμοσμένα στο σημερινό κόσμο. Ε, ε, πρέπει να αναμορφώσουμε το δανειακό σύστημα, το σύστημα χορήγησης δανείων και χορηγήσεων ε, και τα δάνεια θα πρέπει να γίνουν αποτελεσματικά εργαλεία ανάπτυξης. Θέλουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια για να σπρώξουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις και να δημιουργήσουμε καινούριο εργαλείο, καινούρια έννοια ή την συνολική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα είναι ένα, μια πλατιά έννοια που θα περιλαμβάνει όλες τις χρηματοδοτικές ροές. η προϋπόθεση να πετύχουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να μην προσιλωμένη στο στόχο 7. Το θέμα θα ζητηθεί πάρα πολύ φέτος. Ξαναδεσμευτείτε λοιπόν στο σημείο 7 περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια αλλά και πιο εστιασμένη, πιο ευφυής. Μερικά λαμπρά παραδείγματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο με συντηρητικό πρωθυπουργό, ποιο θα το περίμενε αυτό την εποχή της Θάτσερ, έχει αυξήσει κατά 2,7% την ε, ε, αναπτυξιακή βοήθεια σε, στιγμή, σε περίοδο λιτότητας. Οπότε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάνε από μεγάλη λιτότητα, αλλά υπάρχουν και άλλε χώρε που έχουν λιγότερη λιτότητα από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουν αυξήσει την αναπτυξιακή του βοήθεια όσο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στον κύριο Κάμερον. Και τα άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιμηθούν αυτό το παράδειγμα. Τουρκία, άλλο παράδειγμα. Η Τουρκία βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο του ΩΣΑ αυτή τη στιγμή. Και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια κατά από ότι ένας τεράστιος αριθμός ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί το κάνουν αυτό. Ε, ε, είναι παρόμοιος ο λόγος. Ερντοάν και Κάμερον βλέπουν ότι η αναπτυξιακή βοήθεια ε, είναι δείγμα αλληλεγγύης αλλά ταυτόχρονα τη βλέπουν και ως εργαλείο για τις εξωτερικές πολιτικές τους. Ε, θέλουν να δημιουργήσουν αγορέ για τις εταιρείε τους, μακροπρόθεσμα, θέλουν να βοηθήσουν την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, θέλουν να καταπολεμήσουν την ε, ε, λαθρομετανάστευση, θέλουν να σταματήσουν πολέμους, την τρομοκρατία. Η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλα αυτά. Ολοκληρώνοντα να πω ότι λοιπόν ξανά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξαναδεσμευτεί στο σημείο 7 αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συζητήσει και το πώ θα εξυγχρονίσει, θα κάνει πιο ευφυή την αυσιακή βοήθεια. Δεύτερο εργαλείο είναι το φορολογικό. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους μέσω της φορολογίας. Νομίζω ότι εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να μιλάμε πιο ανοιχτά για το ζήτημα αυτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μπορούμε δηλαδή να αυξήσουμε τα έσοδα από τους φόρους έστω και 1% και το οποίο θα μπορούσαμε στη συνέχεια να παρέχουμε προς τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, προς τις χώρες εκείνες οι οποίες χρειάζονται αναπτυξιακή βοήθεια. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω θα καταφέρναμε να διπλασιάσουμε τη συνολική παγκόσμια επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να συλλέξουμε τους φορολογικούς αυτούς πόρους, να καταφέρουμε να τους συγκεντρώσουμε και να αποτελέσουν μια νέα χρηματοδοτική ροή η οποία θα πηγαίνει προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε τις επιδοτήσεις εκείνες οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά. Ο πρόεδρος Γιουκόβε της Ινδονησίας μείωσε τις επιδοτήσεις στα καύσιμα και χρησιμοποίησε το ποσό αυτό όπως οι Νορβηγοί, οι Σουηδοί και οι Λουξεμβουργιανοί προκειμένου να καταφέρουν να βοηθήσουν περισσότερο αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά αυτόν τον τρόπο τα τρία αυτά κράτη χρησιμοποιώντας φορολογικούς μηχανισμούς, φορολογικά εργαλεία, κατάφεραν τελικά να μειώσουν τις επιδοτήσεις τις οποίες δίνανε και κατάφεραν να συγκεντρώσουν περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία δόθηκαν προς αναπτυσσόμενες χώρες με τη μορφή αναπτυξιακής αρρωγής. Νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαν να αντιγραφούν και από άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε και με το φορολογικό τομέα και όντως οι φόροι μπορούν να δημιουργήσουν μια αύξηση των κεφαλαίων εκείνων που δίνονται προς αναπτυσσόμενες χώρες με τη μορφή αναπτυξιακής βοήθειας. Αν δούμε τώρα κάποια αριθμητικά δεδομένα για το τομέα της παιδείας. Πολλές φορές στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι εμείς προωθούμε την ανάπτυξη της παιδείας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα με 2 με 3% του τομέα της παιδείας στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτάται από τη μεταφορά κεφαλαίων και περίπου 99% πληρώνεται τελικά από τους ίδιους τους φορολογούμενους των χωρών αυτών. Δηλαδή οι Βραζιλιάνοι είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν το εκπαιδευτικό του σύστημα, οι Κινέζοι κάνουν το ίδιο, αλλά ακόμα και στην ακτή του λεφαντοστού οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο μέσω της φορολογίας με τη χρηματοδότηση του τομέα της παιδείας. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε εμεί περισσότερο σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η παιδεία, χρησιμοποιώντα κυρίως κάποια φορολογικά εργαλεία. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε μία ομάδα ε, επιθεωρητές στον τομέα της φορολογία χωρί σύνορα, έτσι ονομάζεται η ομάδα αυτή και θεωρώ ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερο στις αναπτυσσόμενε χώρε. Αρρωγή, φόροι και τρίτο τομέα, ιδιωτικέ επενδύσει. Ξέρετε ότι οι ιδιωτικέ επενδύσει μπορούν να συμβάλλουν περί περισσότερο από ότι η επίσημη κρατική αναπτυξιακή αρρωγή. Πολλέ φορέ τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Θεωρώ πάντω ότι το 2015 οι παγκόσμιες επενδύσεις θα είναι περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε 20.000 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό αυτό είναι τεράστιο, είναι ασύλληπτο. Αν συγκρίνεται αυτά τα 20.000 δισεκατομμύρια με τα 150 δισεκατομμύρια που έχουμε συνολικά στα πλαίσια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν να συγκεντρώσουμε όλο και περισσότερα κεφάλαια από ιδιωτικού φορείς αυτή τη φορά, προκειμένου να προωθήσουμε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να διοχετεύσουμε όλο και περισσότερα κεφάλαια σε επενδύσεις στους τομείς αυτούς. Χρησιμοποιούμε λοιπόν και για αυτόν τον τομέα συγκεκριμένα εργαλεία στα πλαίσια της ε, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, προσπαθώντας να μειώσουμε το ρίσκο, τον κίνδυνο που συνδέεται πάρα πολύ, με τις, ε, πάρα πολύ συχνά με, με τις ιδιωτικές επενδύσεις και κατά αυτόν τον τρόπο δίνουμε όλο και περισσότερα κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές. Πολλά αφρικανικά έθνη ουσιαστικά έχουν προσφέρει αυτό το οποίο ονομάζουμε tax holidays, φορολογικές διακοπές για, για πάρα πολλούς ιδιώτες επενδυτές. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε πιο ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες χρειαζόμαστε εμείς ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα ένα νομικό πλαίσιο για τις επενδύσεις αυτές, προκειμένου οι ιδιωτικέ επενδύσει από τη μία χώρα στην άλλη και κυρίω από τον δυτικό κόσμο προ αναπτυσσόμενε χώρε να μπορούν να γίνονται εντελώ νόμιμα και κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο βιώσιμε. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα παγκόσμιο νομικό πλαίσιο για τι ιδιωτικέ επενδύσει στον τομέα τη αναπτυξιακή συνεργασία και τη αναπτυξιακή βοήθεια. Και θεωρώ ότι αν εγκρίνουμε τα νέα αυτά εργαλεία τα οποία σα παρουσίασα θα καταφέρουμε να αυξήσουμε και τι ιδιωτικέ επενδύσει ε, στον τομέα τη αναπτυξιακή βοήθεια. Τέλο. Προσπαθήσαμε από φέτος να προσεγγίσουμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Να καταφέρουμε δηλαδή από κοινού να συνδυάσουμε τόσο το περιβάλλον όσο και την απτυξιακή βοήθεια. Ξέρω ότι θεωρητικά όλοι συμφωνούμε με την προσέγγιση αυτή, αλλά στην πράξη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να συσπυρώσουμε, να συγκεράσουμε, τι δύο αυτέ σχολέ. Αυτή που ήταν υπέρ τη ανεπτυξική βοήθεια για το περιβάλλον και αυτού οι οποίοι προωθούσαν άλλε πτυχέ τη αναπτυξιακή βοήθεια. Προσπαθούμε τώρα να συγκεράσουμε αυτέ τι δύο πτυχέ, αυτέ τι δύο διαστάσει και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμω, πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση και στις δαπάνες, τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία θέλουμε να δώσουμε σε ορισμένες χώρες για επενδύσεις στον περιβαλλοντικό τομέα, μπορούν μόνο να πιάσουν τόπο τελικά αν έχουν και μια έντονη αναπτυξιακή πτυχή. Δεν μπορούμε δηλαδή να χρηματοδοτούμε μόνο περιβαλλοντικές δράσεις. Πρέπει εξ αρχής οι δράσεις μας να είναι τόσο περιβαλλοντικές όσο και αναπτυξιακές. Αυτό θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε και για τα 40 δισεκατομμύρια τα οποία θα πρέπει να δοθούν με τη, μορφή, με τη μορφή ODA, επίσημης αμπτεξικής βοήθειας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει και πάλι εδώ πέρα να έχουμε μια έντονη επίσημη αμπτεξιακή βοήθεια ODA από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όμως να είναι συντονισμένη και να ξέρουμε εξ αρχής ποιο τμήμα των χρημάτων αυτών θα πάει σε περιβαλλοντική δράση και ποιο τμήμα θα έχει να κάνει περισσότερο με αναπτυξιακή βοήθεια. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, Έχουμε τους τρεις αυτούς πόρους, την αρρωγή, τους φόρους και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και στους τρεις αυτούς τομείς χρειαζόμαστε την έντονη συμμετοχή όλων, αλλά θα εξαρτηθεί τελικά από την πολιτική βούληση των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων εταίρων μας για να δούμε αν τελικά θα καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε όλο και περισσότερους ε, ε, πόρους. Ένα 60% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίω προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική σας συμβολή είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά βέβαια πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η συμβολή άλλων μεγάλων κρατών, όπως η Κίνα ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με την κατάλληλη πολιτική βούληση, με το απαραίτητο πολιτικό σθένος, να προωθήσουμε τις επενδύσεις από, όλους, από όλες αυτές τις περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διεξοδική αυτή έκθεση των θεμάτων που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και μια ειδική έκθεση για τα φορολογικά θέματα. Η Έλλη που είναι εδώ το έχει αναλάβει. Ο κύριος Περέιρα έχει να κάνει επίσης ε, με σχετικά θέματα εν ώψη της Αντίσα Μπέμπα και της Συνόδου των Ηνωμένων Με χαρά ακούω ότι πρέπει να ασχοληθούμε και να συσχετίσουμε το θέμα της ανάπτυξης με το περιβάλλον είναι κάτι το οποίο και εγώ ιδιαίτερα έχω υποστηρίξει και πιέζουμε και μέσα στο Κοινοβούλιο να εργαστούμε ως μια ενιαία ομάδα. Άλλωστε η κυρία Μογκυρίνη που θα έρθει να μας ε, μιλήσει σύντομα έχει ηγηθεί της πρωτοβουλίας για, την, ε, για το συγκερασμό μέσα σε μια ενιαία και συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική των πόρων για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Περέιρα που είναι ο συγγητή για τη χρηματοδότηση ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, καλεσμένο μας για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του και για, την, ε, για τις θέσεις που μας εξέθεσε για την ανάπτυξη της ανάπτυξης. Συμφωνώ απολύτως με τη βασική ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να επιβεώσει την στράτευση της για την δέσμευση του 0,7% του ΑΕΠ για την επίσημη ε, κρατική δηλαδή βοήθεια προς την ανάπτυξη. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο γιατί διαφορετικά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ρόλο ηγετικό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα πρέπει το χειτερό δυνατό να προχωρήσει σε αυτό. Θα ήθελα όμως και την άποψή σας σε σχέση με μια παγκόσμια ε, συμφωνία και κατά πόσο θα μπορούσαμε να την περιμένουμε ενώ σε αυτής της διεθνούς διασκέψεως της Αντισαμπέμπα κυρίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη ο κύριος χορηγός σε επίπεδο ενισχύσεων, κρατική αρρωγή. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από τους εταίρους μας ανά τον κόσμο και τι είδους προσδοκίες τρέφει όσα σε σχέση με μια παγκόσμια συμφωνία για το μέλλον της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη από το 2015 και μετά. Και μια δεύτερη ερώτηση σχετική με τους φόρους. Έχετε κάποιους, ε, κάποιες ιδέες, κάποιες παρατηρήσεις σχέση με τη θέσπιση ενός φόρου ...ο οποίος θα απορρέει από τα φορολογικά έσοδα ενός κράτους για να ενισχύσει την ε, ανάπτυξη. Βλέπετε κάτι τέτοιο δυνατό. Και επίσης σε σχέση με τις ιδιωτικές επενδύσεις, αναφερθήκατε στο διεθνές εμπόριο, τι είδου ε, σχέση διαβάζετε μεταξύ διεθνούς εμπορίου και χρηματοδότησης για το εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, έχει επιδοθεί σε μια σειρά από πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ανά τον κόσμο και ρωτώ πώς μπορεί ένα τέτοιο μέσο να αξιοποιηθεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Και μια γενικότερη ερώτηση για τον έλεγχο της δημόσιας βοήθειας, της οποίας το συζητούμε ενώ αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ανησυχούν για το κατά πόσον τα χρήματα που διαθέτουμε φτάνουν εν τέλει στον πραγματικό στόχο. Άρα ερωτώ πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον έλεγχο της αποτελεσματικής χρήσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πάρα από, μια ώρα χρόνο, άρα θα πρότεινα να να ακολουθήσουμε τη διαδικασία ping-pong. Έχουμε τρει σημαντικέ και εκτεθειμένε ερωτήσει. Θέλετε να απαντήσετε πρώτα σε αυτέ, κύριε Σόλχαν, και μετά να ακούσουμε του άλλου. Πολύ ευχαρίστω ε, να απαντήσω ή να ακούσω και άλλε ερωτήσει. Αποφασίστε εσεί. Λοιπόν, κοιτάξτε, εάν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είμαστε και ειλικρινεί, εάν δεν δεσμευτεί για το 0,7% και δεν δεσμεύσει τα αντίστοιχα ποσά, δεν πρόκειται να φέρει αποτελέσματα και θα το δει αυτό μέχρι το τέλο του έτου. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη πολιτική επιλογή. Και πρέπει να προχωρήσει το χειρότερο δυνατόν, να μην χάσει άλλο χρόνο. Λυπή εταίρη, βεβαίω και οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλα εύπορα κράτη πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούν, αλλά πολύ σημαντικό είναι επίσης, πολύ απαραίτητο είναι επίσης να δραστηριοποιηθούν και άλλοι εταίροι, νέα κράτη, η Τουρκία, η Βραζιλία, ναι, ήδη η Κίνα ξέρουμε ότι προσφέρει αναπτυξιακή έρωγη περισσότερο, αλλά και λαμβάνει σε έναν βαθμό. Λοιπόν, έχουμε κράτη τα οποία μετακινούνται σιγά σιγά και θα βρεθούμε σύντομα να βλέπουμε ε, μικρό αριθμό, βασικά Ηνωμένε Πολιτείες Ευρώπη, να είναι καθαρή χορηγή, έναν άλλο μικρό αριθμό κρατών, ε, κυρίως Αφρικής, να είναι μόνο ε, ωφελούμενοι ή δικαιούχοι αυτής της βοήθειας αλλά έναν μεγαλύτερο αριθμό κρατών να βρίσκεται στην διάμεση κατηγορία που και δέχεται και προσφέρει. Γιατί μπορεί να έχει, επί παραδείγματι, ωφεληθεί από τη μεταφορά τεχνολογίας από τη Γερμανία, η Τουρκία, παραδείγματι, αλλά από τη δική της την πλευρά προσφέρει αναπτυξιακή βοήθεια στη Σομαλία ως δε μουσουλμανικό κράτος μπορεί να έρχεται εγκύτερα με τα, με τα κράτη αυτά και να έχει και τη σχετική εμπειρία από την προσφορά αναπτυξιακή βοήθεια. Μπορεί το Μεξικό από την άλλη να λαμβάνει αναπτυξιακή βοήθεια στην, ε, από τις ΗΠΑ αλλά μπορεί να προσφέρει από την πλευρά του αρρωγή σε άλλα κράτη όπως ε, η IT. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι παραδείγματι, τα μένα αλλάζουν στάση πέρυσι. Αυτά δείχνουν πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος. Ε, φόρος, φόρος από, την, από τα δημοσιονομικά έσοδα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασιστεί σε ύψιστο τελικά πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διεθνής κοινό, κοινότητας θα θέλαμε να το δούμε. θα πρέπει όμως να δούμε και πώς στην πραγματικότητα θα υλοποιηθεί γιατί είχε και στο παρελθόν ε, προταθεί ένα συγκεκριμένο φόρος για την ανάπτυξη που όμως στη συνέχεια έχασε τον προσανατολισμό του και χρησιμοποιήθηκε σε άλλες ε, εφαρμογές από τους υπουργούς, ενώ η Γαλλία ήταν μεταξύ των λίγων κρατών που τον διατήρησε ως καθαρά αναπτυξιακό φόρο. Και ναι ε, στο θέμα των συναλλαγών είναι χρήσιμες βεβαίως ε, για την ανάπτυξη, αλλά τα μικρότερα φτωχότερα κράτη δεν μπορούν να ωφεληθούν από αυτές, όσο ελεύθερες και να συναλλαγές αν επισκεφθεί κανείς την Ορβηγία στο σούπερ μάρκετ, δεν θα βρει πάνω από μισό της εκατό προϊόντων προερχομένων από την Αφρική. Όχι γιατί υπάρχουν ε, ε φραγμοί στο εμπόριο, αλλά γιατί δεν μπορούν ε, τα αφρικανικά κράτη να διατηρήσουν μια αλυσίδα προμήθειας, παραγωγής και προμήθειας, που να ε, οδηγεί τα προϊόντα της στο, στις ξένες αγορές. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πωλήσει ακατέργαστες πρώτες ύλε, αλλά τίποτε άλλο. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι προπτικές είναι θετικές για την Κίνα, για την Τουρκία και άλλες χώρες της Ασίας που μπορεί να μεταφέρουν τους χώρους παραγωγής τους στην Αφρική και να αναπτύσσουν έτσι συστήματα εμπορικά με, την, ε, με τις χώρες αυτές, Αιθιοπία, Σενεγάλη, Ρουάντα, επίσης έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον. Επίσης, όταν ήμουν υπουργό ε, στη Νορβηγία, όλο και πιο συχνά μου έλεγαν το εξής. Σε παρακαλώ, Μέρεκ, πήγαινε να επισκέπτεσαι τις φτωχές χώρες Αφρικής για να βοηθάς τους ανθρώπους. Και πρέπει να ξέρουμε ότι τα χρήματα που διαθέτουμε δεν είναι χρήματα που καταλήγουν στις τσέπες κάποιων δικτατόρων, αιμοσταγών. Είτε, τα, είτε προσφέρουμε τον έρανό μας στην εκκλησία για να τον διοχετεύσει τη φτωχή αφρικανική χώρα, είτε μέσω ενός φόρου αναπτυξιακού, θέλουμε να ξέρουμε πάντα τα λεφτά αυτά. Και μπορεί να είναι μεν δαπανηρό ή να περιπλέκει λίγο και να καθιστά λιγότερο αποτελεσματική την αξιοποίηση αυτής της βοήθειας. Πρέπει να έχουμε συστήματα όσο το δυνατόν πιο στεγανά για την καταπολέμηση της διαφθοράς τους αναπτυξιακούς σπόρους. Ασφαλώς δεν μπορούμε να την εξαλείψουμε 100%. Αλλά μέσα σε ένα σύστημα όπως υπάρχει ε, πρέπει να κάνουμε το μέγιστο δυνατό για τον περιορισμό της διαφθοράς και της καταστρατήγησης των πόρων. Επίσης ε, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ε, χαρακτηριστικό το ότι λόγω της διαφθοράς αυτής παραμένουν στη φτώχεια και την ένδυα τόσοι πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ ο Γκάβο που έχει την ε, έκθεση για την περίοδο μετά το 2015. Ευχαριστούμε πολύ για όλες, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Με το ψήφισμα μας το Νοέμβριο ε, εκφράσαμε τη δική μας άποψη που είναι πολύ συμπίπτη με τη δική σας ε, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το σημείο 7 είναι ένα από τα κέρια σημεία. Το Κοινοβούλιο επιμένει σε αυτό το θέμα εδώ και καιρό. Σε ό,τι δεν αφορά την διαφθορά και τις παράνομες δωρές κεφαλαίων, το είπατε κι εσείς ε, ότι ε, το ποσό των παράνομων ροών που βγαίνει από τις ανεπτυγμένες χώρες και φτάνει στις ανεπτυγμένες χώρες υπερβαίνει κατά πολύ την αναπτυξιακή βοήθεια που δέχονται αυτές τις χώρες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. θα πρέπει να το συζητήσουμε με την Κομισιόν. Ο κ. Μίμητσα κάποια στιγμή είχε υποσχεθεί να δει το θέμα αυτό και να δει αν μπορεί η Κομισιόν να κάνει κάτι. Θα πρέπει πάντως να το εξετάσουμε. Και αυτό με φέρνει και στο ζήτημα της σημασίας των ε, ε, θεσμικών οργάνων που δεν αποκλείουν κανέναν. Στο ανακοινωθέν της Επιτροπής Αμψιακής Βοήθειας υπάρχει ένα σημείο που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Θα, το ερώτημα μου το εξή. Σε αυτό το ανακοινωθέν λέει ότι ε, συμφωνούμε να δια, πώς μπορούμε να λάβουμε αυτό το θέμα υπόψη μας. Ίσως να το αντιμετωπίσετε εν μέρη με την συνολική ε, με την έννοια της συνολικής αναψυχιακής βοήθειας ε, θα μας απαντήσετε όμως. Είπατε επίσης ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες αναπτύσσονται και ταυτόχρονα αυξάνουν την και τους βοήθεια, αλλά, υπάρχουν, αλλά αυτές οι χώρες πολύ συχνά είναι χώρες οι οποίες υποχωρούν σε ό,τι αφορά το θεσμικό κομμάτι τους, ε, την, ε, τη δημιουργία θεσμικών οργάνων χωρίς ε, αποκλεισμούς. Πώς μπορούμε, να, μπορούμε να, αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. <coughs> On, on the first one, I mean, there is Στο πρώτο θέμα, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες ροές κεφαλαίων στον κόσμο θα πρέπει να μειωθούν και έτσι κι αλλιώς επιμένουμε για τη διαφάνεια σε όλους τους τομείς. Οι φορολογούμενοι μας ε, ζητούν ότι θέλουν να ξέρουν τα πάντα για την προσωπική ζωή των πολιτικών για παράδειγμα και το ίδιο κάνουν και τα μέσα με τις ενημέρωσης. Ταυτόχρονα ε, επιτρέπουμε ένα τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας να περνάει από φορολογικούς παραδείσους με βασικό στόχο να κρυφτούν. Ακόμα και αν δεν, είναι παράνομα, δεν έχουν αποκτηθεί παράνομα πολλοί, περνούν από τους ε, φορολογικούς παραδείσους για να κρύψουν τον ε, ιδιοκτήτη τους. Ε, η Νορβηγία το 1990 είχε ένα τύχημα, το μεγαλύτερο τύχημα της ιστορίας της, 200 άτομα πέθαναν σε, σε ένα τάνκερ το οποίο πήρε φωτιά ε, και 20 χρόνια μετά ακόμα δεν ξέρουμε σίγουρα ποιος ήταν πάνω σε αυτό το πλοίο. Συγγνώμη, δεν ξέρουμε ακόμα σίγουρα σε ποιον ανήκε το πλοίο. Ε, δεν έχουμε καταφέρει να αποδώσουμε ευθύνες και να αποδώσουμε δικαιοσύνη. πώς είναι δυνατόν ο καπιταλισμός να είναι υπεύθυνο αν επιτρέπει τέτοιου είδους σχήματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ένας πρόσκαμικών του της Ενωμένου Βασιλείου είπε ότι η Starbucks, η Google και η Microsoft, τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του, των Πολιτειών δεν πληρώνουν φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, είναι πιθανό να πληρώνουν στον ΕΠΑΛ το τον Ισημερινό Αλλά δεν πληρώνω στον Βασίλειο. Καταλαβαίνετε ποια είναι η προφανής απάντηση. Οπότε ο ΣΑ έχει ξεκινήσει ε, την προσπάθεια ε, να καταπολεμήσει την ε, διάβρωση φορολογικής ε, βάσης και τις παράνομες ροές κεφαλαίων. Δεν ε, θέλουμε να γίνονται μετακινήσεις ε, κεφαλαίων για αποφυγή της φορολογίας. Η αυτόματη ε, ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού τύπου, για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει. Αυτό όμως είναι πιο εύκολο μεταξύ ανεπτυγμένων χωρών. Ίσως είναι πιο δύσκολο όμως να λειτουργήσει στη Γουινέα Μπισάου για παράδειγμα γιατί δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να υποστηρίξει ένα τέτοιο σύστημα. Οπότε θα πρέπει να βοηθήσουμε τα ανεπτυσσόμενες χώρες να χτίσουν καλύτερα φορολογικά συστήματα. Το άλλο ζήτημα που θέτεται είναι ίσως ακόμα πιο δυσεπίλητο. Σίγουρα είναι πολύ πολιτικό. Κατά η άποψη δική μου άποψη είναι εξή. Οι success stories της ε, ανάπτυξης δεν έγιναν ποτέ σε δικτατορικά καθεστώτα όπως η Βόρεια Κορέα. Ε, ίσως όμως σε αυταρχικά συστήματα όπως η Κίνα. Ναι. Η, Κίν, ε, ε, η Ρουάντα είναι μια άλλη τεράστια επιτυχία από αναπτυσιακής πλευράς αλλά είναι σαφές off the record ότι ο... ότι δεν είναι πραγματική ε, πλήρης δημοκρατία. Έχουμε πολύ λιγότερα παιδιά που πεθαίνουν στον κόσμο από ασθένειες, αλλά και έχουμε τεράστια πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην έχουμε ε, ε, δικαιώματα για ανάπτυξη μιας αντιπολίτευσης σε όλες τις χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Ε, οπότε, ε, όλα τα δικαιώματα θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα. Τα ατομικά, τα κοινωνικο τα εργατικά, όλα τα δικαιώματα μετρούν το ίδιο έχουν την ίδια αξία. Οπότε θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα, αλλά κάθε φορά θα πρέπει οι αποφάσεις μας να λαμβάνονται ad hoc, αναλύοντας την κάθε περίπτωση. Η Σιγκαπούρη είναι πολύ επιτυχημένη χώρα, ε, αλλά από το 1950 και μετά είναι το ίδιο κόμμα στην κυβέρνηση. Ελισάινεν που είναι ε, η συγγήτρια, με συγχωρείτε, για τα φορολογικά ζητήματα τα οποία θίξαμε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Σολχάιμ για την ε, παρουσίαση που έκανε. Είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δυναμώσουμε το φορολογικό καθεστώς που ισχύει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ξέρουμε ότι ο ΣΑ έχει δει ότι κάθε δολάριο το οποίο χρησιμοποιείται ή επενδύεται για τη δημιουργία ενό στεναρού φορολογικού καθεστώτος μπορεί να οδηγήσει σε 650 δολάρια όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα στη συνέχεια. Τι όμως μπορούμε να κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα τυποποιημένο διεθνές φορολογικό σύστημα το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης το σύστημα υποβολής αναφορών αναχώρα όπως γίνεται αυτή τη στιγμή για το τραπεζικό τομέα ή για το βιομηχανικό τομέα, θα πρέπει να επεκταθεί και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, θα πρέπει να καλύπτει και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδίω αν θέλουμε να αποφύγουμε φαινόμενα όπως η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις παράνομες ροές κεφαλαίων, το αναφέρατε και, εσείς στην παρουσίασή σας και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις φορολογικές αρχές των κρατών. Αν γίνει κάτι τέτοιο, πώς μπορούμε όμως να πείσουμε και τις απτυσσόμενες χώρες να συμμετέχουν. Έχουμε προβλήματα εδώ, το είπατε κι εσείς. Πολύ συχνά δεν έχουν τα απαραίτητα θεσμικά όργανα προκειμένου να υποβάλουν τέτοιες πληροφορίες. Δεν υπάρχει απαραίτητη υποδομή. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να καταφέρουμε κατά κάποιο τρόπο να ενισχύσουμε τις δομές των κρατών εκείνων ώστε να μπορούν να μας παρέχουν και αναπτυσσόμενες χώρες τις απαραίτητες φορολογικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όντως έχουμε εγκρίνει αυτή τη στιγμή κάποια εργαλεία τα οποία για παράδειγμα αφορούν τις τράπεζες οι οποίες μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για κεφάλαια τα οποία έχουν ε, χρησιμοποιηθεί παράνομα και οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να διοχετεύονται περισσότερο ή να ανταλλάσσονται ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναπτυγμένες χώρες. Η Σουηδική κυβέρνηση, για παράδειγμα, θα ήταν πολύ σημαντικό σε επαφές που έχει με τις χώρες στις οποίες βοηθά να μπορεί να έχει ως συνομιλητή, ως αξιόπιστο συνομιλητή μια φορολογική αρχή στην απτυσσόμενη χώρα η οποία να λειτουργεί σωστά. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά έχουμε φορολογικέ αρχέ στην απτυσσόμενη χώρε υποστελεχωμένε με ανθρώπου που δεν έχουν το κατάλληλο επίπεδο για να επιτελέσουν το έργο το οποίο καλούνται να κάνουν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την δημιουργία τέτοιων στεναρών αξιόπιστων φορολογικών δομών στις απτυσσόμενη χώρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει βέβαια μία νυχτή, αλλά υπάρχουν πολλές σχετικές πρωτοβουλίες από διάφορες χώρες. Η Νορβηγία για παράδειγμα, η ομάδα στην οποία αναφέρθηκα, επιθεωρητές στο φορολογικό τομέα χωρίς σύνορα, είναι φορεί που έχουν υποβάλει τέτοιε σχετικέ πρωτοβουλίε. Όπω είπατε κι εσεί πάντω, η πρωτοβουλία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί όντω μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να επενδύσουμε μέσω του φορολογικού τομέα σημαντικά ποσά τα οποία θα έχουν και μια πάρα πολύ σημαντική απόδοση στη συνέχεια. Μπορούν να λειτουργήσουν δηλαδή πολλαπλασιαστικά. Όσον αφορά αυτή την αναχώρη υποβολή αναφορών, νομίζω ότι το εργαλείο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σαφώ δεν θα πρέπει να γίνει ένα γραφειοκρατικό εργαλείο, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει άχθος. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι χρήματα καταβάλει μία επιχείρηση σε μία συγκεκριμένη χώρα, για παράδειγμα στην Αφρική. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η οικονομική δραστηριότητα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης στην Αγγόλα ή σε οποιαδήποτε άλλη αφρικανική χώρα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να επεκταθεί όμως το σύστημα αυτό και σε άλλους τομείς έτσι ώστε όλες αυτές οι πληροφορίες να είναι πλέον ξεκάθαρες, να μην υπάρχει απόκρυψη πληροφοριών. Ο Νέσ έχει το λόγο, ο αντιπρόεδρο μα, ο οποίος όμως είναι και εισηγητή για τα ζητήματα αντιξιακή βοήθειας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια και την έκκληση υποστήριξη προ τη Σρι Λάνκα. Ξέρω πόσο σκληρά εργαστήκατε όλα αυτά τα χρόνια, την τελευταία 20 ετία, για να βοηθήσετε στην επάνωδο της ειρήνης στη Σιλάνκα. Ενώ κάποιοι αμφισβητούσαν και τη δουλειά σας και την, το κύρο σας και τις καλές σας προθέσεις επειδή δεν ήθελαν την ειρήνη αλλά τον πόλεμο στη Σιλάνκα. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να είστε υποψήφιος και για τον Νόμπελ Ειρήνης. Σας συγχαίρω για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει στην προσπάθεια για την επάνωδο της σε αυτό το μικρό νησί. Αυτό που θέλω να σα ρωτήσω. Έχει να κάνει με τις εξωδικαιικές δραστηριότητες αναπτυσσομένων κρατών. Γιατί είχα μια σχετική έκθεση εγώ στο Κοινοβούλιο που για πρώτη φορά ομόφωνα ε, υιοθετήθηκε. Αφορούσε τα ε, δικαιώματα ιδιοκτησίας. και εκεί έκανα σαν αφήγηση το εξή υπόθεση. Έλεγα στο κείμενο δώστε ένα κομμάτι γης με τους πρόσφυγες όλου του κόσμου και θα μπορέσω μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να ετοιμάσω ένα κράτος ευημερούν. Έτσι λοιπόν, και γιατί γίνεται αυτό, διότι και το είδαμε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουμε έναν τρόπο ανάπτυξης πλούτου έχουμε κόσμο σε ε, περιοχές στα φτωχά αυτά κράτη οι οποίες είναι παραγκουμπόλεις μέσα όμως σε πλούσιες περιοχές στη Βομβάη παραδείγματι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε, σε, ε, σε ακριβά κομμάτια γης αλλά δεν έχουν τίτλους, δεν έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας και δεν καταγράφονται επίσημα, δεν έχουν αξία στα χέρια τους, καμία οικονομική αξία και αν θέλουν να πουλήσουν ένα κομμάτι γης ή μια παράγκα, την πουλάνε σε ένα φίλο τους, με όποιους όρους, χωρίς όμως επίσημους τίτλους, χωρίς ε, βιβλία, καταστατικά ε, από και το καθεξής. Έχουμε να κάνουμε μια τεράστια αξία σε δισεκατομμύρια, μη καταγεγραμμένη λοιπόν. Μπορούμε να κοιτάξουμε το θέμα αυτό πιο προσεκτικά. Απάντηση. Ναι, ξέρω ότι υπάρχει μια κίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο με τον Ντεσότο επικεφαλή τον οικονομολόγο από το Περού, για την αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των φτωχών να είναι πιο εύκολο δηλαδή να εξασφαλίσουν δάνεια, να ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση και να είναι και πιο δύσκολο οι κρατικές αρχές ή κάποιοι πλούσιοι με επιρροή να τους πετούν στο δρόμο. Ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να εξασφαλιστεί. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές στον κόσμο όπου οι ισχυροί μπορούν να πετάξουν στο δρόμο ανθρώπους που έχουν ζήσει εκεί γενναίες γεννών χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Κάποιες χώρες έχουν αντιμετωπίσει με πιο ικανοποιητικό τρόπο από ό,τι άλλες τα ζητήματα. Παραδείγματι στην Κίνα υπάρχουν καλύτερα συστήματα αποζημίωσης σε περίπτωση όπου ε, αναγκαστικά μετακινούνται για λόγους ανάπτυξης. Για το νέο αεροδρόμιο του Πεκίνου, παραδείγματι, θα χρειαστεί η μετακίνηση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Ε, έχει θεσπιστεί ένα σύστημα υποστήριξης, ε, βοήθειας και αποζημιώσεων, το οποίο φαίνεται να δουλεύει αρκετά καλά. Και μάλιστα βλέπουμε κάποιους να πηγαίνουν Προβλέποντα ότι μπορεί να ενταχθεί σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο μια περιοχή και άρα θα γίνουν οι απαλωτριώσει σχετικέ, και να αγοράζουν και η γη περιμένοντα τη σχετική αποζημίωση από την απαλωτρίωση. Άρα μπορεί και πρέπει το κράτο να αναλαμβάνει αυτή την δέσμευση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, Πρόεδρο της Επιτροπής ε, για την Αναπτυξιακή Βοήθεια. Θα ήθελα ωστόσο να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις και ανησυχίες η οποία είναι η εξή, η οποία είναι η εξής, ότι νομίζω δεν αναγνώσουμε σωστά την κατάσταση όπως έχει. Πριν από 20 χρόνια οι φτωχοί βρισκόταν αποκλειστικά στι αναπτυσσόμενε χώρες. Τώρα η πλειονότητα των φτωχών βρίσκεται στις ε, αναδυόμενε χώρες. Ε, παλιότερα τις βλέπαμε στις ε, άκρες των δρόμων στο Γουαγκαντούγκου, στην Κινσάσα, εκεί που έμπαινε ο δρόμος στην πόλη. Βλέπαμε ανθρώπους που μπορεί να βγάζανε 5 cents την ημέρα και να παραμένουν ακόμα στις χώρες αυτές, σε αναδυόμενες όμως χώρες, οι φτωχοί απλώς φορτώνονται σε λεωφορεία και απομακρύνονται για να μην ενοχλούν τους επισκέπτες, τους ξένους επισκέπτες. Γιατί λοιπόν ε, δεν ξεκαθαρίζει ένα μήνυμα ε, ως προς την ανάγνωση κατάσταση και όσα ενόψη της βέβαια. Θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα γεγονότα αυτά να τα καταγγείλουμε, να καταπολεμήσουμε την φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις αναδυόμενες. Είπατε ότι υπάρχει επαρκής παραγωγή πλούτου και πόρων σε αναδυόμενες ε, χώρες ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Αλλά δεν μοιράζεται, δεν κατανέμεται σωστά αυτός ο πλούτος. Άρα, εάν κοιτάξουμε πιο πολύ εις βάθος, και επιδιώξουμε μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της ένδυας, πρέπει να αναστήσουμε τις πηγές της ένδυας. Διαφορετικά θα έχουμε χάσει μια πολύ σημαντική ευκαιρία σε αυτό το έτος που έχει χαρακτηριστεί, έχει ονομαστεί και έτος κατά της, ε, υπέρ της ανάπτυξης. Επίσης τα 150 δισεκατομμύρια για την αναπτυξιακή βοήθεια για το για την ανάπτυξη, κυρίως για την ε, καταπολέμηση της φτώχειας. Φοβούμε ότι αυτά τα 150 δισεκατομμύρια θα χαθούν κατακαιρματιζόμενα σε μικροδράσεις για το ένα και το άλλο θέμα, λίγο κλιματική αλλαγή, λίγο ε, καταπολέμηση από εδώ, αλλά μεγάλα ζητήματα όπως αυτό του ιού του έμπολα δεν θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Και είπα τον έμπολα γιατί είναι μεν μολυσματική νόσος, είναι λοιμώδης νόσος, αλλά δεν επεκτείνεται λόγω της, ε, του ιού. Επεκτείνεται γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα εγκαίρως. Γιατί έχουμε να κάνουμε περιοχές που έχουν πληγεί από εμφύλιο πόλεμο από χρόνια τώρα και που δεν έχουν προχωρήσει σε διαρθρωτικές προσαρμογές. Και από τη Σύνοδο της Ουάσιγκτον που έχουμε κάνει λάθος επιλογές ε, συνεχίζουμε και αντί να αντιμετωπίζουμε συστημικά τις κρίσεις ε, περιοριζόμαστε σε επιφανειακές μόνο παρηγορητικές ε, ρυθμίσεις κάνουμε πολύ λίγα και με μεγάλη καθυστέρηση όπως και με την, οικονομική, με την χρηματοοικονομική κρίση αν θέλουμε λοιπόν το έτος αυτό για την ανάπτυξη να καταστεί χρήσιμο πρέπει να έχουμε μια πιο εντός εισαγωγικών επιθετική στάση μια πιο αποφασιστική δηλαδή στάση και εσείς όσα έχετε τη δυνατότητα ε, και τα πρακτικά μέσα να εμπλακείται σε εσωτερικά ζητήματα των κρατών. Για τα φορολογικά είναι, για, για το σύστημα της παιδείας είναι, μπορείτε και εφόσον οι επικρίσεις σας αφορούν τους πάντες, δεν μπορείτε να κατηγορηθείτε και για διακριτική μεταχείριση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια επιλεκτική στάση, πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη στάση και αυτό όχι μόνο ως κράτη, γιατί αναφέρεστε στα κράτη για την ανάπτυξη, αλλά ερωτώ πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των πολλών αυτών φτωχών που υπάρχουν στα αναδυόμενα κράτη τους οποίους αγνοούμε ουσιαστικά γιατί αναδυόμενον το κράτος θεωρεί ότι δεν χρειάζεται πια να ασχοληθεί με τους φτωχούς του. Δεν είναι α, α, ε, ε, θέμα αλληλεγγύης διεθνούς κατά πολέμηση της φτώχειας. Γιατί ξαφνικά γίνεται ζήτημα εσωτερικής ε, πολιτικής. Τι θα πούμε για τα αναδυόμενα κράτη σαν τη Σεντεβέμπα. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ πιο οξύ στην ρητορική μας, να δώσουμε λύσεις αποτελεσματικές. Ιδάλλως σε 10-15 χρόνια θα καλούμε πάλι σε μια νέα σύνοδο με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως τα λέμε και πάλι, αλλά θα είναι αποτυχημένη η θα προσπαθούμε να καλύψουμε χαμένο έδαφος. Πάντως, εάν τα ίδια αίτια προξενούν τα ίδια αποτελέσματα, θα πρέπει να αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, ε, μιλήσατε για την συνέντευξη της Ουάσιγκτον. Τίνουμε να ξεχνάμε πόσο καταστροφικός ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Όχι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ήταν ε, κατά βάση ε, επιτυχία. Ε, σε σχέση με το, την καταστροφή που είχε στην υπόσταση υπόλοιπο κόσμο. Για δύο λόγους. ε, όλοι οι ε, βάρβαροι δικτάτορες του κόσμου υποστηρίχθηκαν είτε από το ένα στρατόπεδο είτε από το άλλο. Ε, με το επιχείρημα ότι είναι κτίνος αλλά είναι το δικό μας κτίνος. Ε, και μετά ε, υπερβολική απελευθέρωση των αγορών στην ε, Δύση οδήγησε σε αρνητικές αντιδράσεις με ακρότες προς την άλλη κατεύθυνση. Ε, και η απόλυτη απελευθέρωση και η απόλυτη κεντροσχεδιασμένη οικονομία ήταν άκρα τα οποία πέτυχαν και γι' αυτό λόγο μετά τον ψυχρό πόλεμο πετυχαίνουμε πολύ περισσότερο. Ε, σχεδόν όλοι στον κόσμο προωθούν μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση. Ένα κοινωνικό κράτος με ελεύθερες αγορές. Αυτό έχει αποδειχθεί πολύ πιο επιτυχημένο από ότι η σοβιετική ιδεολογία ή η υπερβολική, α, ε, υπερβολικά φιλελεύθερη οικονομία. Τώρα, Πού είναι η φτώχεια. Ε, στις αναδυόμενες ή στις ανεπτυσσόμενες χώρες. Ε, πολλοί πιστεύουν ότι η στις ανεπτυσσομενες χωρες πολλοι πιστευουν οτι η κινα θα φτάσει στη μηδενική φτώχεια. Ε, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στη Λατινική Αμερική. Ε, οπότε οι αναδυόμενες χώρες έχουν κάνει πάρα πολλά βήματα. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Η φτώχεια μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα. αλλά κυρίως ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Ε, έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 10% κάτι που έχει οδηγήσει σε ε, πάρα πολύ μείωση της ε, φτώχειας. Βέβαια, εμείς είχαμε πει ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε κρυζώσει τη φτώχεια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με οικονομική ανάπτυξη. Σε καμία περίπτωση ακόμα και η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας να οδηγήσει στην απόλυτη κρύωση της φτώχειας στην Αφρική για παράδειγμα. Πρέπει στην ανάπτυξη ε, να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. ποιε είναι οι πολιτικές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν στην πραγματική εκρίζωση της ακραία στόχιας. Η ανάπτυξη είναι χρήσιμη βέβαια, χρειάζεται η ανάπτυξη, αλλά πρέπει να έχουμε και άλλες πολιτικές. Για παράδειγμα, ε, δωρεάν ενίσχυση ε, των πιο φτωχών τμήματων του πληθυσμού, πέτυχε στη Λατινική Αμερική, μικροπιστώσεις, ε, συνταξιοδοτικά, καινούργια συνταξιοδοτικά συστήματα, όπως βλέπουμε στην Ινδονησία. Και άλλα εργαλεία έχουμε. για να καταπολεμήσουμε την ακραία φτώχεια. Έχουμε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες ε, περισσότερο κόσμο στην υπεθροπότη της ότι ε, και, και μεγάλο κύμα του πληθυσμού μακριά από τα πολιτικά κέντρα. Ε, με βάση αυτό το, το πανόραμα θα πρέπει να εστιάσουμε τις πολιτικές μας. Thanks. Um, Lola Θα είμαι λίγο πιο τεχνική σε ό,τι αφορά τα νέα μέτρα που έχουν εγκριθεί. Ε, εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να δημιουργηθεί μια καινούρια μέθοδος ε, υπολογισμού των ε, πιστώσεων, των δωρεάν πιστώσεων. Υπάρχουν όμως κάποια δικά και πια αρνητικά. Σε ό,τι αφορά τα θετικά, πολύ σωστά που θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις ε, καθαρές ροές βοήθειας και την βιωσιμότητα του χρέους ως κριτήριο για την χορήγηση ενισχύσεων. Σε ορισμένα σημεία θα μπορούσαμε να πάει λίγο ακόμη πιο μακριά, όπως για παράδειγμα το ποσοστό αναφοράς ε, των, ε, της δωρεάν, των δωρεάν πιστώσεων που ε, ε έμεινε στο 10%. Ε, το, ΑΕ, το Διεθνές Ταμείο συνδέει αυτό το δίκτυο με το αμερικανικό δολάριο και αυτό δεν είναι σωστό. Θα έπρεπε ε, να δούμε και ποιο είναι το κόστος για τον ε, δέκτη βοήθειας, για να δεχτεί αυτή τη βοήθεια. Μετά έχουμε ε, ένα ελάχιστο ποσοστό ερεσιμότητας που συνδέεται με το μέσο εισόδημα. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τις χώρες που έχουν μικρότερα εισοδήματα που όμως εξακολουθούν να έχουν ανάγκες ενίσχυσης. Τώρα, στα αρνητικά. Ε, δεν είναι σωστό που έχει, ίδιο, έχει ε, εισαχθεί ένας ε, διορθωτής, διορθωτικός παράγοντας με βάση τον κίνδυνο διότι δεν λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος αυτού που δέχεται τη βοήθεια του λήπτη. Επίσης, δημιουργούνται προβλήματα σε ό,τι αφορά την, την διαγραφή του χρέους. Τούτου ε, τούτο λεχθέντος είναι σημαντικό να, ε, να, δούμε ότι ενδεχομένως δεν θα πρέπει να εστιάσουμε τη βοήθεια στις πιστώσεις. Από την αρχή της κρίσης οι δωρεάν πιστώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί ε, σαν να είναι αναπτυξιακή βοήθεια γιατί θεωρείται ότι μπορεί να επιστραφεί. Επίσης οι δωρητές δεν θα πρέπει να προσπαθούν προσπαθούν ε, να χρησιμοποιούν μόνο ε, πιστώσεις ε, διότι αυτό δημιουργεί προβλήματα χρέους, υπερβολικού χρέους. Τι, θέλω να πείτε τι πιστεύετε για όλα αυτά, αλλά η πιο βασική μου ερώτηση είναι θα υποστηρίζατε την πρόταση το 85% της ενίσχυσης να είναι δωρεάν και να μην στηριζόμαστε τόσο πολύ στις πιστώσεις. Θα μπορούσατε, πιστεύετε, αυτό να γίνει υποχρέωση. <clears throat> Πάρα πολλά σημαντικά σχόλια και επικρίσεις για τον συμβασμό του Δεκεμβρίου. Ε, όλοι οι πολιτικοί συμβασμοί ε, έχουν αυτό το αρνητικό γιατί έχουν είναι πολλές οι, οι απόψεις και κανένας συμβασμός δεν είναι τέλειος. Κανένας συμβασμός όλη την ιστορία και πολύ περισσότερο στη Σρι Λάγκα για παράδειγμα δεν ήταν τέλειος. Όμως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι πριν το συμβασμό. Παραδείγματα. Παλιότερα ε, ε δεν γινόταν διάκριση ανάμεσα στα ε, δωρεάν ε, δάνεια και στα, μη ε, ανάμεσα επιδοτούμενα και μη επιδοτούμενα δάνεια. Τώρα γίνεται η διάκριση και είναι λογικό. Παλιότερα είτε κάποιο έδινε ένα δάνειο στη Βραζιλία, την Κίνα ή την Τουρκία, είτε το έδινε στην Τανζανία, τη Μοζαβίκη και το Μαλάουι, ε, ήταν το ίδιο πράγμα. Τώρα ε, υπάρχει μια προτίμηση για δάνεια σε λιγότερο αναπτυγμένε χώρε με συγκεκριμένες βέβαια όρου όρους ε, για τη δημιουργία, του, ε, δημιουργία προς του χρέου. Τώρα, ε, η δωρεάν ενίσχυση πράγματι πολλέ φορέ είναι προτιμότερη από τα δάνεια. Γι' αυτό το λόγο και η δωρεάν βοήθεια είναι πολύ ψηλότερη σε αναπτυσσόμενες χώρε από ότι τα δάνεια. Αλλά και τα δάνεια έχουν να παίξουν το ρόλο τους η, τα δάνεια ε, θα παίξουν, πρέπει να παίξουν σημαντικότερο ρόλο για τις χώρε χώρες που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα. Επίσης μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην ε, δημιουργία ε, υποδομών, αυτοκινητοδρόμων κλπ. Παρά βέβαια σε άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση, υγεία κλπ. Οπότε είναι και τα δύο εργαλεία. Ο συμβιβασμός ε, πιστεύω δεν ήταν σίγουρα τέλειος, αλλά είναι ένα τεράστιο θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο δεν ε, δέχθηκε και πολλές κριτικές. ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Γαλλία και η Γερμανία ε, και η Απωνία δευτερευόντως ε, χορηγούν το μεγαλύτερο αριθμό δανείων. Ε, τα ιαπωνικά δάνεια είναι και πιο χαλαρά μάλιστα σε ό,τι αφορά τους όρους τους. Ε, κυρίως όμως η Γαλλία, η Γερμανία και, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί που χορηγούν τα περισσότερα δάνεια. Ε, οι άλλε χώρε έχουν και πολύ αστερότερου όρου όπω η Σουηδία, η Νορβηγία ή και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα έρθει σήμερα το απόγευμα εδώ και θα μα εξηγήσει το ε, σύστημά τη ε, για τη χορήγηση δανείων. Είναι ο κύριος Φαν Μπάλεκομ. Um, Κυρία Χαουτάλα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο που βλέπουμε ότι εσείς ως επικεφαλής Επιτροπής Μεταξυξής Βοήθειας του ΩΣΑ πραγματικά συμβάλλετε πάρα πολύ στην αναθεώρηση, την επικαιροποίηση της προσέγγισης που έχουμε για την δεξιακή βοήθεια. Οι τρεις άξονες που αναφέρατε, συνδρομή, αρρωγή, φόροι και ιδιωτικές επενδύσεις, είναι όντως πάρα πολύ σημαντικοί. Και αν δεν κάνω λάθος η DAC έλαβε πρόσφατα κάποιες αποφάσεις όσον αφορά την ODA, την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ισχύει ότι ε, η DAC ε, δεν έθεσε συγκεκριμένο ποσοστό του ODA που θα πρέπει να ισχύει για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και αν ναι για ποιο λόγο λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ενδεχομένως τα άλλα μέσα ανάπτυξης να είναι πιο χρήσιμα, να είναι πιο ωφέλιμα για τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες. Επίσης, όσον αφορά την TOSD, τη συνολική επίσημη υποστήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την νέα αυτή έννοια την οποία αναφέρεται, νομίζω ότι δεν θα αντικαταστήσει την ODA, αλλά θα συμπληρώσει την επίσημη αντιξιακή βοήθεια, έτσι δεν είναι. Ελπίζω ότι μέσω του νέου αυτού μέσου δεν θα προσπαθήσουν κάποιες χώρες να μειώσουν το ποσοστό τους ODA, το ποσοστό επίσημης αντεξιακής βοήθειας. Όσον αφορά τώρα το φορολογικό τομέα, σας ευχαριστώ για την προσωπική σας δέσμευση. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εσείς, και το είπατε κι άλλος το ίδιος, ήσασταν αυτός που ξεκίνησε το σύστημα αυτό των Tax Inspectors Without Borders φορολογικοί επιθεωρητέ χωρί σύνορα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που έχετε καταβάλει προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στα φορολογικά καθεστώτα των αναπτυσσομένων χωρών. Όσον αφορά τώρα τι ιδιωτικέ επενδύσει, νομίζω ότι εδώ πέρα πάλι ακούσαμε κάποιε πολλά υποσχόμενε ιδέε. Θα μπορούσατε να μα μιλήσετε λίγο για το ζήτημα του impact investment, δηλαδή τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι επενδύσει ή μπορείτε επίση να αναφερθείτε περισσότερο στη δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους πιο φτωχούς στις πιο φτωχές χώρες και τέλος πάλι στην αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις. Μα είπατε ότι χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Αναφερθήκατε στην προστασία των επενδυτών επίσης. Επομένως, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία δίκαιη συμφωνία όσον αφορά κάποιους συγκεκριμένου επενδυτικούς κανόνες θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε μια τέτοια συμφωνία. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει και την Επιτροπή μας και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια του TTIP νομίζω ότι δεν λαμβάνουμε αρκετά υπόψη μας τις επιπτώσεις μιας τέτοιας μελλοντικής ενδεχόμενης συμφωνίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας άποψη όσον αφορά αυτό το νομικό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Απάντηση. Προφανώς υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχουν ζητήματα με το νομικό αυτό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το παράδειγμα διαφόρων επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται και βρίσκονται σε θέση ισχύω κάθε φορά που διαπραγματεύονται με μια κυβέρνηση και στη συνέχεια μπορεί να προκύψει μια νέα κυβέρνηση στην απτυσσόμενη χώρα η οποία ενδεχομένω να θέλει να προχωρήσει σε νέε διαπραγματεύσει. Κάτι τέτοιο θα συνέβαινε ούτω ή άλλω και σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να το αποφύγουμε, να παραπονεθούμε για το ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι να δούμε αν πραγματικά σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει ένα πραγματικό σφαιρικό νομικό πλαίσιο για τη διευθέτηση προβλημάτων, συγκρούσεων ανάμεσα σε μία επιχείρηση ή μία κυβέρνηση, αν προκύψουν δηλαδή προβλήματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ορισμένε χώρε βλέπουμε ότι υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τι επιχειρήσει για του δικού του κομματικού ε, λόγου ή πολλέ φορέ ακόμα και για να πλουτίσουν οι ίδιοι. Επομένω, όταν μια μεγάλη επιχείρηση επενδύει σε μια προβληματική χώρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το νομικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκα. Δεν καλύπτει αυτό τόσο πολύ κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες πολύ προσωρινά και βραχυπρόθεσμα δραστηριοποιούνται σε μια χώρα αναφέρομαι περισσότερο στις μεγάλες εκείνες επιχειρήσεις οι οποίες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επιθυμούν να επενδύσουν σε μια απτυσσόμενη χώρα. Οι ίδιες αυτές οι επιχειρήσεις απαιτούν και ζητούν αυτό το σταθερό νομικό πλαίσιο. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές φορές κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες αισθάνονται ότι είναι κάπως απομονωμένες στην όλη αυτή η συζήτηση, ότι βρίσκονται απλώς αντιμέτωπες με τους πολιτικούς ηθήνοντες, με εμά από την άλλη πλευρά, χωρίς όμως να ξέρουν σε ποιο πλαίσιο τελικά κινούνται. Στα πλαίσια του νομικού αυτού πλαισίου θα έχουμε έναν συντονισμένο συνεχή τέτοιο διάλογο, σε επαφές που είχαν πρόσφατα Κινέζοι με μια Σουηδή, Σουηδική τράπεζα είπαν όντω ότι χρειάζονται αυτό το συνεχή διάλογο προκειμένου να καταφέρουν να επιλύουν προβλήματα τα οποία ενδεχομένω να προκύπτουν. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι το μέσο αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις. Όσον αφορά το, την έννοια του impact investment, αυτό νομίζω ότι πολύ συχνά το συγχαίουμε με τη φιλανθρωπία, όπου πολύ συχνά απλώς χορηγούμε, δίνουμε χρήματα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό όμως δεν είναι impact investment. Η έννοια του impact investment έχει να κάνει με μια επένδυση που κάνει κάποιος σε μια χώρα, από την οποία όμως περιμένει κάτι σε επιστροφή, περιμένει μια απόδοση. Δηλαδή πρόκειται για στοχευμένη επένδυση για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Για παράδειγμα, ένα καλύτερο σύστημα ε, περιβαλλοντικές υπηρεσίες περιβαλλοντικέ υπηρεσίε καθεξής. Χρειαζόμαστε περισσότερο τέτοιο impact investment, Κυρίως ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερες, μάλλον λιγότερες πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες που συμβάλλουν στο impact investment, ενώ από την άλλη έχουμε την Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συμβάλλουν αρκετά σε αυτό το μέσο επένδυσης. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο ακόμα για τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να επενδύουν περισσότερο ακόμα και να προχωρούν σε κάποιες φιλανθρωπικές δράσεις. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να σκεφτούμε το παράδειγμα του Bill Gates ή κάποιον άλλων σημαντικών επιχειρηματιών που συμβάλλουν πάρα πολύ σε αυτού του είδου την ανθρωπιστική αρρωγή. Νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα θα έπρεπε να βλέπουμε όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη δικαιολογία ότι πληρώνουμε υψηλότερου φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τους 8 πιο πλούσιους ε, ανθρώπους στον κόσμο, των οποίων το εισόδημα αντιστοιχεί στα χρήματα τα οποία διαθέτουν ε, τα 3,5 εκατομμύρια πιο φτωχοί άνθρωποι στον κόσμο. Έχουμε έναν φορέα, ένα ταμείο στην Νορβηγία, το οποίο συμβάλλει σε αυτόν τον τύπο της επένδυσης ε, πάρα πολύ, ε, κάνει πάρα πολλές φιλανθρωπικές δωρές. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει η Νορβηγία να έρθει σε επαφή με κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημιουργήσουν οι χώρες αυτές από κοινού ένα ταμείο Impact Investment. Δεν λέμε ότι θα πρέπει τα χρήματα αυτά να δοθούν δωρεάν σε κάποιες χώρες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο το οποίο θα έχει τη μορφή επενδυτικού ταμείου. Ένα, 1% μόνο των χρημάτων αυτών που θα μπορούσαν να δοθούν μέσω τέτοιων ταμείων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πάρα πολύ μεγάλη απόδοση των επενδύσεων αυτών, Ιδίω στην εποχή αυτή που βλέπουμε ότι μειώνται τόσο πολύ οι τιμέ των καυσίμων. Τέλος, η έννοια αυτή τη συνολική επίσημη υποστήριξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το TOSD, είναι ένα νέο λοιπόν μέσο το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ζητήματα όχι μόνο αναπτυξιακής βοήθειας αλλά και ζητήματα εγκαθίδρυσης της ε, ειρήνης, διατήρησης της ειρήνης ή της ασφάλειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ένα ποσοστό του ταμείου αυτού, του μέσου μάλλον αυτού του χρηματοδοτικού θα μπορούσε να δοθεί και για τέτοιες ε, δράσεις. Νομίζω ότι ε, Πρέπει εμεί να είμαστε σε θέση μέσω τη αναπτυξιακή βοήθεια σε χώρε όπω η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για παράδειγμα, να προωθούμε και το ζήτημα τη ασφάλεια. Τέλο, χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Το είπατε κι εσεί αυτό. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου ένα 50% τη αναπτυξιακή βοήθεια θα πηγαίνει όντω στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Δεν αναφέρομαι βέβαια στο 50% του ODA κάθε χώρα ξεχωριστά. Και αυτό γιατί κάθε χώρα συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο. Αν δούμε την Ευρώπη, για παράδειγμα, η, Πολωνία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, οι οποίε ε, αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει να δίνουν επίσημα αναπτυξιακή βοήθεια, έχουν δικά του προγράμματα τα οποία βοηθούν βαλκανικέ χώρε, βοηθούν την Μόλδοβα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, ιστορικέ πολλέ φορέ φιλικέ σχέσει μεταξύ συγκεκριμένων κρατών Επομένως υπάρχουν χώρε οι οποίε υποστηρίζουν συγκεκριμένε χώρε. Δεν υπάρχουν ε, πολλές χώρε οι οποίε μέσω επίσημης αντικειμενικής βοήθειας υποστηρίζουν για παράδειγμα την Μόλδοβα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι με την προώθηση των λιγότερων απτυγμένων χωρών θα σταματήσουν ε, οι χώρε αυτέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθούν τη Μόλδοβα. Επίσης η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία επιθυμούν να παρέχουν επίσημη ανεπτυξιακή βοήθεια κυρίως στις Φιλιππίνες, στην Ινδονησία ή σε κάποια μικρά νησιωτικά κράτη του ειρηνικού. Αυτό είναι απόλυτα λογικό. Και προφανώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν πρόκειται να παρέχουν ODA σε μικρά νησιωτικά κράτη του ειρηνικού. Όταν λοιπόν λέω 50% του ODA δεν αναφέρομαι ε, ξεχωριστά σε κάθε κράτος, αλλά το 50% συνόλου της επίσημης αντιξιακής βοήθειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέρινεν τώρα, πρώτος από τους τρεις επόμενους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Έρικ, για την παρουσία σας και για τις απαντήσεις. Συμφωνώ, όπως ξέρεις, με τις βασικές ιδέες που εκφράζεις. Δεν είναι τυχαίο που εκπροσωπεί την Νορβηγία από σένα και από την ε, Κρόπρου Χάρλεμ ε, στον τομέα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, αναπτυξιακής βοήθειας που ξεκίνησε από το δεκαετία του 80. Έχω δύο ερωτήσεις καταρχάς σχετικά με το εμπόριο. Ο γύρος της Ντόχα στον ΠΟΕ ξεκίνησε ως γύρος αναπτυξιακός με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης μέσω του διεθνούς εμπορίου. Υπήρξαν δυσκολίε βάσει των οποίων εξασφαλίστηκε μια κάποια λύση τώρα, αλλά εγώ ανησυχώ ιδιαίτερω για τις συνέπειες της συμφωνίας TTIP διατλητικού εμπορίου με τις ΗΠΑ Πολιτείες που προχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνίες οι οποίες διαβρώνουν τη βάση για μια Παγκόσμια Εμπορική Συμφωνία ευνοϊκή για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, Ερικ, πόσο μεγάλο κίνδυνο βλέπει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα έπρεπε να κάνει για να αποτρέψει τέτοιου είδου δυσμενεί εξελίξει. Επίση, ε, ο ΣΑ και η Αναπτυξιακή Επιτροπή είναι σε διεθνή διάλογο, σε διαρκή διάλογο με δωρητέ. έστω και αν δεν είναι ακόμη μέλη. Πώς μπορούμε λοιπόν να καλέσουμε τους δωρητές να ακολουθήσουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε τους δραστηριότητα. Έχεις δει κάποιες θετικές εξελίξεις προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Φερρυπίν ε, κάποια αλλαγή στις πολιτικές ε, επιλογές της Κίνας ή άλλων νέων δωρητών. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ Πάουλ. με χαρά μιλάω με Φιλανδούς είχαμε πάντα πάρα πολύ καλές σχέσεις και ιδιαίτερα στο τομέα της ανάπτυξης δεν έχει θέση όμως η Επιτροπή ούτε εγώ ιδιαίτερες γνώσεις για το θέμα των ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων ίσως να χαρακτηριστούν από τον ΠΟΕ ε, κάποια στάδια που θα οδηγούσαν σε μια γενικότερη εμπορική συμφωνία, παγκόσμια εμπορική συμφωνία ή ως εμπόδια. Πάντως είναι προτιμότερες ε, εμπορικές συμφωνίες που θα συμπεριλαμβάνουν και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πάντως για τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες το πρόβλημα δεν είναι η απουσία συμφωνιών ή η ύπαρξη εμποδίων στο εμπόριο. Άλλα είναι τα προβλήματά τους. Και έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με την Ορβηγία που θέλησε να βοηθήσει στην ε, κατάσταση ε, σφαγίων με βάση κάποιες προδιαγραφές στην Ουγγάντα. Οι περιορισμοί λοιπόν ε, που προέκυψαν ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ζώα τα οποία θα μπορούσαν να σφαγιαστούν με βάση κτηνιατρικούς και υγειονομικούς κανόνες. Χρειαζόταν μια ζώνη αποκλεισμού, για ένα-δύο εκατομμύρια κεφάλια ε, γύρω από το σφαγείο με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες γεωνομικούς και εκτινιατρικούς που θα ε, εμπόδιζαν τον, την επιμόλυνση και αυτό δυσκόλεψε πολύ τα ζητήματα. Αυτό βέβαια την πρόοδο στο θέμα αυτών των σφαγείων. Αυτό βέβαια μπορεί να θεωρηθεί από τον τοπιο πληθυσμό ως εμπορικό εμπόδιο αλλά για μας ήταν ζήτημα προστασίας του πληθυσμού και βέβαια ε, εξασφάλισης της αποδοχής και για τους Ευρωπαίους. Μετά υπήρχε ζήτημα μεταφορών. Ε, δεν υπάρχουν ε, θαλάσσιες μεταφορές που να μπορούν να εξασφαλίσουν μια πρόσκοπτη μεταφορά προς το λιμάνι και από το λιμάνι των σφαγίων. Είναι λοιπόν τα συνοδευτικά προβλήματα. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε συναλλαγές με την Κίνα παρά με την Αφρική αυτή τη στιγμή για διάφορου τέτοιου λόγους. Αλλά ασφαλώ πρέπει να συζητηθεί το θέμα του εμπορίου για τους δωρητές. Είναι βεβαίω πολύ σημαντικό το να έχουμε κύριες και πέραν των ευρωπαϊκών κρατών ω κύριες ομάδες δωρητών τους Άραβες και τους Κινέζους όπως τώρα συμβαίνει και άλλους δωρητές βεβαίως έχουμε όπως η Βραζιλία αλλά δεν προσφέρει η Βραζιλία τόσο υψηλά ποσά. Άραβες και Κινέζοι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην πρώτη θέση από πλευράς Αράβων. Περιμένουμε και το Κατάρ να ενισχύσει την συνδρομή του και βέβαια συνεργαζόμαστε όλο και πιο στενά με την Κίνα. Θα πρέπει πιστεύουμε να απορρίψουμε την ιδέα που επικρατεί τόσο πολύ στην Ευρώπη ότι ό,τι κάνει η Ευρώπη είναι υπέροχο και ότι ό,τι κάνει η Κίνα δεν είναι τόσο καλό. Ε, νομίζω ότι πρέπει να επωφεληθούμε και από τα όσα κάνει η Κίνα. Πολλά είναι τα προβλήματα βεβαίως εκεί. Κάποιε είναι οι εταιρείε οι οποίες ε, δεν δρούν σωστά στο αναπτυξιακή δράση τους, ε, ευρωπαϊκές εταιρείες σε παραδείγματι, οι οποίες φέρουν τους δικούς τους ε, Κινέζους δηλαδή εργάτες να δουλέψουν όταν αναλαμβάνουν κάποιο έργο στην ε, Αφρική. Από την άλλη όμως οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν χτίσει ούτε ένα κομμάτι δρόμου στην Αφρική. Ενώ οι Κινέζοι κάνουν ε, κάποιες προσπάθειες αναπτυξιακές ε, στις διάφορες περιοχές της Αιθιοπίας, της Ερυθρέας και άλλο. Και επίσης από την άλλη έχουμε ειδικού οι οποίοι πηγαίνουν στις χώρες αυτές από την Ευρώπη και δεν μένουν στα Χίλτον και τα λοιπά, γιατί και αυτό ενοχλεί φυσικά στα ακριβά ξενοδοχεία, αλλά σε καταβλισμούς και σε παράγκες και από την άλλη έχουμε Κινέζους οι οποίοι όταν πηγαίνουν εκεί έχουν το δικό τους φαγητό και όλο τον εξοπλισμό όπως τον θέλουν και δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα. Δεν είμαστε όμως πια στην κατάσταση που ε, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είμαστε οι μόνοι ε, χορηγοί βοήθειας ή οι μόνοι καλοί χορηγοί βοήθειας. Το ίδιο ισχύει για μας όπως για τους Κινέζους Αμερικανούς. Υφιστάμεθα επικρίσεις για διάφορους λόγους και είναι καλό να γίνεται η συζήτηση και να ενισχύεται η προσπάθεια. Θες να συμπληρώσεις κάτι, αλλά πολύ σύντομα, σε παρακαλώ, 20 δευτερόλεπτα. Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν το δυναμικό τους μέσω της ενίσχυσης για το εμπόριο. Επίσης ε, περιέγραψες μη δασμολογικούς φραγμούς νομίζω. Έρικ, πρέπει και αυτοί να αντιμετωπίζονται στις εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μία σύντομη ερώτηση για τη χρηματοδότηση η επαλλαγή από το χρέος ή η η αναδιαταξη χρέους έχει καμία σημασία για σας στην αξιολόγησή σας αυτής της ε, βοήθειας. Έχουμε παραδείγματι ε, ποσά που έχουν καταβληθεί για την ενίσχυση τομέα της υγείας, περιπίν. Ε, επίσης έχω μια ερώτηση, Γραμμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι συνδυάζονται επιτέλους το περιβάλλον με την ανάπτυξη. Είπατε σε ιδιώτες επενδυτές ότι θα πρέπει και αυτοί να κινητοποιηθούν και να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους σε πράσινους στόχους. Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι μπορούν να κινητοποιηθούν αυτοί οι ιδιώτες ε, επενδυτές και τι είδους κοινωνικές προδιαγραφές μπορεί να υπάρχουν ή τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ε, αμέσως. Ευχαριστώ όλα αυτά τα πολύ ξεκάθαρα παραδείγματα που μας δίδεται ιδιαίτερα. Να δούμε λίγο το σχόλιο σας όμως, ότι σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, ή, μάλλον το γεγονός ότι ε, η φτώχεια κινείται από τις αναψώμενες χώρες στις αναδυόμενες χώρες. Πώς γίνεται αυτό, αφού μια χώρα γίνεται πιο πλούσια Πώς γίνεται η φτώχεια να ακολουθεί. Ε, λέμε ότι για να μην έκανε την απόλυτη φτώχεια χρειάζεται ένα δολάριο τη μέρα. Στη Γερμανία ο, το ημερομίσθιο είναι 8,5 ευρώ ε, την ώρα. Ε, ποια, ποιοι είναι οι κανόνες λοιπόν για να καθορίσουμε το τι είναι το ελάχιστο. Ε, Πώς και θεωρούμε ότι μια χώρα είναι αναδυόμενη και όχι αναπτυσσόμενη πια. Ε, χρησιμοποιείται μακροοικονομικά μεγέθη μόνο ή μεγέθη που με την καθημερινή ζωή. Start ναι, πολύ κρίσιμα αυτά τα θέματα. Ο ορισμός της φτώχειας, απόλυτη φτώχειας είναι το 1,25 δολάρια ανά ημέρα και ανά άτομο είναι ο, ο, ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Να δούμε και όλους τους άλλους ορισμούς, αλλά δεν θα ήθελα να αλλάξουμε αυτόν τον ορισμό γιατί είναι αποδεκτός από όλους. Αυτό είναι, ε, αυτός είναι ο παγκόσμιο αποδεκτός ορισμός. Τώρα, ε, η φτώχεια έχει σχέση και με την ενέργεια, με το περιβάλλον, με τα καθημερινά έξοδα και το πώς αυτά διακυμαίνονται κλπ. Σίγουρα. Τώρα, το αν ένα κράτος είναι αναδυόμενο ή αναπτυσσόμενο, δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει ορισμός. Το, η κάθε χώρα αυτό ορίζεται ως το ένα ή το άλλο οι αναδυόμενες αγορές, είναι, οι χώρες είναι κυρίως Βραζιλία, Κίνα ε, και Ινδία. Ινδία. Ε, τώρα, η ανάπτυξη διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ε, τώρα, η όλη η Νοτιοανατολική Ασία είναι μεγάλη επιτυχία σε ό,τι αφορά τη φτώχεια. Το ίδιο και στη Λατινική Αμερική. Η Βολιβία ήταν η χώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και μετά το Περού σε ό,τι αφορά τη φτώχεια. Αλλά παντού ήταν επιτυχής η ανάπτυξη στην ε, ε, Λατινική Αμερική. Η Κολομβία είναι αυτή τη στιγμή τη μόνη πολιτική στρατιωτική εκκρεμότητα που υπάρχει σε όλη την Ήπειρο, Βόρεια και Νότια Αμερική. Όμω, σε ορισμένα κομμάτια τη Αφρική, ίσω από τη Γουινέα Μπισάου μέχρι τη Σομαλία και στη Μέση Ανατολή και στην Νότιο Ασία υπάρχουν ακόμα εκκρεμή προβλήματα. Θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν εκεί. Ε, και εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Παγκόσμια Τράπεζα. Κύριε Χόιμπακ. Ένας τρόπος να προωθήσουμε τις πράσινες επενδύσεις ε, είναι η αναπτυξιακή βοήθεια να αναλάβει το πρόσθετο κόστος, αν υπάρχει προς το κόστος για την προώθηση των αναλλακτικών μορφών ενέργειας. εναλλακτικό έναντι των ορυκτών υδρών αθράκων. Εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, αναπτυξιακή βοήθεια με πάρα πολλού τρόπου και να την συνδυάσουμε με ιδιωτικέ επενδύσει, να πάρουμε τον κίνδυνο τη ιδιωτική επενδύση και να τον καλύψουμε με την αναπτυξιακή βοήθεια. Για παράδειγμα, όταν δεν υπάρχει ένα σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια χώρα, είναι πολύ δύσκολο ε, να εγκαταστήσουμε ε, φωτοβολταϊκά. Οπότε ενδεχομένω θα μπορούσαμε εκεί να χρησιμοποιήσουμε την αναψυχιακή βοήθεια. Η μεγάλη αποτυχία ε, θα ήταν να τα αφήσουμε όλα αυτά στις αγορές. Και αυτό έχει γίνει το δεκαετία του 80. Λέγαμε, δεδομένου ότι εμπορικά οι ε, ανακτικές μορφές ενέργειας ε, είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις, να το αφήσουμε στις αγορές όμως. Αφήνοντα τι αγορέ, δεν δημιουργήθηκε ένα υδροελεκτρικό σταθμό παραγωγή ενέργεια στην Αφρική. Οπότε τώρα έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Η, αυτό που έχει κάνει η Γερμανία είναι παράδειγμα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, έχει τεράστιο δυναμικό και έχει και τεχνογνωσία. Ε, άλλωστε έχουν πέσει τόσο πολύ τα κόστα της, ε, το, κόστη των φωτοβολταϊκών που είναι εναλλακτική λύση σε πολλά μέρη του κόσμου. Η ελάφρυνση του χρέους είναι και αυτή ένα εργαλείο αλλά γενικά το χρέο αυτή τη στιγμή δεν είναι υπερβολικά βαρύ σαν τι επόμενε χώρε. Μιανμάρ για παράδειγμα. Έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση που έχει ανοίξει τον κόσμο, προωθεί τι οικονομικέ αλλαγέ, προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα με τι μειονότητε. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε εδώ και τέσσερι δεκαετίε θα έπρεπε αυτή η κυβέρνηση να πληρώνει τα χρέη τα οποία είχαν συσσωρεύσει οι προηγούμενες στρατιωτικές κυβερνήσεις και με τόκους και χρεολύσια για δάνεια τα οποία είχαν συναφθεί το 1970 το, το, 80 αστρονομικά ποσά τα οποία έχουν συσσωρευτεί αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να υποχρεωθεί η καινούργια κυβέρνηση να τα πληρώσει. Ε, Καμία κυβέρνηση θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορεί εύκολα κανεί να, ε, δεν θα μπορούσαν να να έχουν πρόσβαση σε αγορές και σε καινούργια δάνεια αν δεν κάνουν κάτι και για το χρέο. Οπότε, ναι, θα πρέπει να ελαφρυνθεί το χρέο, αλλά ταυτόχρονα να αποφύγουμε ε, οι χώρε να ξαναγυρίσουν σε υψηλά επίπεδα χρέου μετά. Επίσης δεν θα πρέπει να προωθούμε και να δίνουμε κίνητρα σε ανεύθυνο δανεισμό. Στην Νορβηγία, ας πούμε, ναι, δώσαμε ελάφρυνση χρέου σε πολλές χώρες για χρέη τα οποία είχαν συσσωρευτεί προκειμένου να προωθήσουμε την αφηγική μας βιομηχανία. Και όταν τη δεκαετία του 1980 δεκαετία 80 και δεκαετία του 90 είχαμε πρώτα την αφηγική μας βιομηχανία. Προσπαθήσαμε σε χώρες όπως το Περού, η Σημερινός κλπ. να ε, δανείσουμε ε, μεγάλα τεράστια ποσά για να προωθήσουμε την αφηγή μας βιομηχανία, ποσά τα οποία αργότερα δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν. Okay, well, I think Mr. Solheim has given us... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σολχάιμ ε, έκανε πολύ σκληρή προσπάθεια, μας παρουσίασε πάρα πολλά θέματα. δύο ώρες περίπου με ερωτήσεις και απαντήσεις. Ελπίζω να σας ταλαιπωρήσουμε πολύ. Πάντως είδαμε θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα ε, για τις επενδύσεις, για τον δυτικό τομέα, για τα φορολογικά ε, εν γέννη για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Διακόψουμε για λίγο για να έρθει η επόμενη ομιλήτρια εκ μέρους της Λετωνική Προεδρίας. Okay, colleagues, if people could take their seats. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξανακαθίσουμε σας παρακαλώ θερμά για να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. I think you can sit next to the minister. You have staff here. Okay, colleagues, we're going... Αγαπητοί συνάδελφοι, με χαρά καλωσορίζω σήμερα την κυρία Καλενιά Λουκατσεβίκα, Υπουργό για τα Ευρωπαϊκά Θέματα της Λετωνίας, παρακολουθεί εκ του συνέγγυ το έργο της Επιτροπής μας και τις σημερινές παρατηρήσεις θα τις εστιάσει κυρίω σε θέματα απτώμενα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναφέραμε και νωρίτερα ότι κηρύχθηκε έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους για την ανάπτυξη στη Ρήγα πριν από 10 μέρες περίπου. Πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Πρέπει όμως και να σημειώσω ότι και η ιδέα για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης προήλθε από λετονικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που το ζήτησαν και έτσι με χαρά είδα την, ε, στην εκδήλωση αυτή στη Ρήγα τις ε, προσπάθειες, τις στράτες στην αποφασιστικότητα και της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό παρόντα για να κηρύξει την έναρξη του Ευρωπαϊκού έτους. Αλλά και εσείς ξέρω ότι είσαστε ε, αποφασισμένοι να ε, εξασφαλίσετε την επιτυχία αυτού του Ευρωπαϊκού έτους. Με χαρά σας βλέπω λοιπόν εδώ σήμερα. Στον ανθρωπιστικό τομέα έχουμε πολλές προκλήσεις Έχουμε έκθεση για το θέμα της επέκτασης ε, και της έδωσης του ιού του έμπολα, γιατί τι συνέβη, τι πήγε στραβά, τι δεν έγινε σωστά. Έχουμε να κάνουμε την ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν, γιατί στο Νότιο Σουδάν, όπως και βέβαια τη Συρία, το Ιράκ, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Γάζα, έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Μεγάλα λοιπόν ζητήματα και θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας παρέμβαση και τις ιδέες σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με χαρά έρχομαι σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και την παρουσία σας στη Ρήγα πριν από μερικές μέρες. Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι λοιπόν εδώ με μεγάλη χαρά για να συστήσουμε τα σχέδια και τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πριν όμως προχωρήσω στις προτεραιότητες και την παρουσίασή τους, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Ιταλική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διασφάλισαν την ε, απρόσκοπτη μετάβαση στο νέο κύκλο της Λετωνικής Προεδρίας. Πρέπει πιστεύω να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε να δώσουμε περισσότερη ενεργητικότητα στο έργο της Ένωσης και να το καταστήσουμε πιο ορατό για τον πολίτη. Έχουμε λοιπόν εστιάσει σε τρία θέματα, την ανταγωνιστικότητα, την ψηφιακή οικονομία και τη στράτευση της Ευρώπης στις προτεραιότητες μας, θέματα που νομίζω αφορούν όλους τους Ευρωπαίους. Έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντικές οικονομικές, γεωπολιτικές, στρατηγικές και σε επίπεδο ασφαλείας πολύ σημαντικές αλλαγές. Έχουμε προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε. Η Ένωση μπορεί να προσφέρει μεγάλη δυνατότητα για δράση μεγάλη ποικιλία επιλογών. Όμως εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουμε την απόφαση για τη λήψη δράση και διασφάλιση των αξιών μας. Δεν υπάρχει λοιπόν νομίζω καλύτερο τρόπος να επιδειχθεί η παγκόσμια στάδευση της Ευρώπης από την ε, βοήθεια την αρρωγή που προσφέρουμε στους πιο ευάλωτους της περιοχές κρίσεως ανά τον κόσμο. Άρα λοιπόν σήμερα θέλω να αναφερθώ σε τέσσερις προτεραιότητες για τη λετωνική προεδρία στο χώρο της ανθρωπιστικής, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντιμετώπιση κρίσεων, προαγωγή ανθρωπιστικών αξιών, ανάπτυξη και προετοιμασία της Ανθρωπιστικής Συνόδου του 2016. Πρώτο λοιπόν καθήκον μας, ε, στο ανθρωπιστικό μας θεματολόγιο είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται ταχαίω και με συμπόνια στι ανθρωπιστικέ κρίσει. Αυτό δεν είναι απλή υπόθεση γιατί ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια ανά τον κόσμο δεν φαίνεται να συρρυκνούνται το αντίθετο μάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερι κρίσει επίπεδου τρία Και αυτό είναι το ύψιστο επίπεδο κατεπήγοντο με βάση την κατάταξη των ΗΠΑ. Στη Συρία, το Ιράκ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά και στο Νότιο Σουδάν. Έχουμε επιπλέον μια επιδημία έμπολα με καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς της Γουινέας, της Λιβερίας, της Ιεραλαιώνα. Αυτά όμως είναι η πιο, το πιο ορατό κομμάτι των προκλήσεων. Πολλές άλλες ανθρωπιστικές κρίσεις και ανάγκες προκύπτουν από φυσικές καταστροφές ή καταστροφές που ξενεί ο άνθρωπος, απολυσμονημένες κρίσεις, Παραδείγματι στην Ιεμένη έχουμε, πάνω από, έχουμε σχεδόν 15 εκατομμύρια ανθρώπους που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Η Λετωνική Προεδρία λοιπόν θα συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος του τρίου μεταξύ Ιταλίας, Λετωνίας, Λουξεμβούργου και μέσω του ρόλου μας ως προεδρεύοντος στο Συμβούλιο ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια και την επιστηστική βοήθεια, το ΚΟΧΑΦΑ ε, και τη σχετική ομάδα εργασίας θα προαγάγουμε στρατηγικό συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και επιτροπή. Στόχο μα είναι η συλλογική ανταπόκριση Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ανθρωπιστικέ κρίσει να είναι στο δυνατόν πιο αποτελεσματική και ταχεία. Ταυτόχρονα όμω η Λετωνική Προεδρία ε, θα εξασφαλίσει και ότι δεν θα λησμονηθούν οι λησμονισμένε ε, κρίσει από το ε, χρονοδιάγραμμα των εργασιών του Συμβουλίου Κοχάφα προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη για τις συνεχιζόμενες ανάγκες ε, για προσφορά αρρωγής και, σε άλλες, ε, και άλλες δράσεις. Δεν πρόκειται να υπησαλθώ σε λεπτομέρειε σχέση με την ε, ανάγκη για τα απόψη Ευρωπαϊκής Ένωση σε συγκεκριμένε καταστάσεις ανθρωπιστικών κρίσεων, αλλά υπάρχουν κάποιε τι οποίε οπωσδήποτε θα πρέπει να εκθέσω διεξοδικότερα. Η Σύρια ασφαλώς είναι μια είναι η κρίση με την κατεξοχή ε, μεγαλύτερη εμβέλεια σε θέματα ανθρωπιστικά αλλά και ασφάλειας έχουν ξεπεράσει το όριο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της ως αρρωγή από την αρχή της κρίσης συνεχίσουμε την προσφορά αρρωγής προς όλες τις χώρες που άμεσα ή πιο άμεσα επηρεάζονται από την κρίση η Προεδρία λοιπόν θα εξασφαλίσει και ενισχύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ε, στην εξέταση, την αξιολόγηση του πώς μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην υλοποίηση της έκκλησης των Ηνωμένων Εθνών του Δεκεμβρίου, αν θα χρειαστεί δηλαδή μια νέα διάσκεψη χορηγών και αν θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε συντονισμό προκαταβολικά μεταξύ κρατών μελών και επιτροπής. Επίσης η επιδημία του ιού έμπολα είναι μια άλλη κρίση που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Έχει φέρει τεράστιες καταστροφές στη Γουινέα, τη Λιβερία, τη Σιεραλεόνε. έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την ε, συγκεντρωτική, μια, μια συλλογική ανταπόκριση έχουν αρχίσει να δίνουν αποτελέσματα. Υπάρχει μια ενίσχυση και επιτάχυνση της αρρωγής, προσαρμογή σε μια ε, μεταβαλλόμενη διαρκώς κατάσταση υπό την καθοδήγηση του Επιτρόπου Στυλιανίδη ο συντονιστή για την ε, ανταπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδημία του έμπολα. Τώρα πρέπει να διατηρηθούν οι δεσμεύσεις και το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν υποσχεθεί τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εκταμιευθούν ταχύτατα και αποτελεσματικά. Κύριος στόχος κατά τη Λετωνική Προεδρία θα είναι η προαγωγή της, ε, του αναλογισμού σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας επιδημίας σε ολόκληρη τη Δυτικοαφρικανική περιοχή. Η Προεδρία ιδιαίτερα υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ΙΣΥΠΑ της Εκπροσώπου και της Επιτροπής για την Οργάνωση μιας μεγάλης, μιας ευρείας διεθνούς διασκέψεως το Μάρτιο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα μακροπρόθεσμα ζητήματα. Και θα ήθελα να αναφερθώ με λίγα λόγια και στην Ουκρανία. τα δεινά που περνάει ο κόσμος εκεί τα βλέπουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία και στη χώρα μου και έτσι υποστηρίζουμε και θεωρούμε πρόσδεκτη την ενίσχυση της ανθρωπιστικής ε, αρρωγής αλλά και της πολιτικής προστασίας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το στρατηγικό σχέδιο ανταπόκριση 2015 των Ηνωμένων Εθνών ως Προεδρία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την επάνωδο στην ε, ειρήνη και τη σταθερότητα. Κύριε και κύριοι βουλευτές, ε, στόχος μας επίσης είναι η τήρηση των τέσσερων ανθρωπιστικών αρχών της ανθρωπιάς, ουδετερότητας, αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. Πρόκειται για αρχές οι οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Θα καθοδηγηθούμε σε όλες μας τις δράσεις από την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, όπως έχει συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Καλωσορίζουμε τα αποτελέσματα της ε, περσινής αξιολόγησης της συνένεσης αυτής. Προτεραιότητα δε της Λετωνικής Προεδρίας είναι να εξασφαλίσει χώρο για εις βάθος συζήτηση των συμπερασμάτων και συστάσεων αυτής της αξιολόγησης. Πρέπει η συζήτηση δε να συνοδευτεί από συγκεκριμένε δράσεις. Η Λετωνική Προεδρία θα προσπαθήσει να ενισχύσει την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ακούγεται όλο και πιο δυνατά η φωνή της ανθρωπιάς και του ανθρωπισμού. Παράλληλα θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το σεβασμό για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την πρόσβαση ε, στην, στην αρρωγή των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη. Ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις αρχές μπορεί να προσφέρεται και πρέπει να προσφέρεται μόνο όπου υπάρχει εξασφάλιση και της ε, ασφάλειας των, ανθρωπιστικών, των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό χώρο και του ιατρικού προσωπικού. Έχουμε ε, φαινόμενα όπως η απαγωγή ε, εργαζομένων στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας αυτήν την εβδομάδα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που μας υπενθυμίζουν με τρόπο επώδυνο τους κίνδυνους. Θέλουμε επίση να συνεχίσουμε την προστασία γυναικών και κοριτσιών σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη. Απλά μέτρα όπω η βελτίωση του σχεδιασμού των καταπλησμών προσφύγων η διαχείριση ασφάλειας μπορούν να φέρουν τεράστια βελτίωση. Κυρίε και κύριοι, ο τρίτος τομέας που θέλω να υπογραμμίσω σήμερα σχετίζεται με την ανακούφιση και την ανάπτυξη και την προαγωγή της ε, διατήρησης αυτής της υποστήριξης. Όπως ήδη δήλωσα, η Λετωνική Προεδρία θέλει να εξασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική αρρωγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών παραμένει ανεξάρτητη, χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι θα έχουμε επαφέ μεταξύ των δικών μας, ε, του δικού μα ανθρωπιστικού και άλλων ε, παραγόντων. Πρέπει να υπάρξει κοινή ανάλυση και ε, διεξοδική επισκόπηση των αναγκών για να έχουμε και ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ιδιαίτερα υπάρχει ανάγκη για εταιρική σχέση μεταξύ ανθρωπιστικών ε, ειδικών αλλά και ειδικών στην ανάπτυξη, ώστε η αποκατάσταση και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη να σχεδιάζονται για να εξασφαλίσουν διάρκεια, αντοχή. Η καλύτερη ανοικοδόμηση, οικοδομούμε με καλύτερο τρόπο, είναι απαραίτητη για να περιοριστεί ο κίνδυνος μελλοντικών καταστροφών. Δεν μπορούμε δηλαδή να συνεχίσουμε να δαπανούμε σε μεγάλη κλίμακα ποσά για ανθρωπιστική βοήθεια σε επανερχόμενους διαρκώς φυσικούς ε, κινδύνους και καταστροφές. Προάγει λοιπόν η Λετωνική Προεδρία την καταγραφή της αντοχής των ευρωπαϊκών στρατηγικών. Αναθεωρούμε όπου υπάρχει ανάγκη με βάση το σχέδιο δράσεως για την αντοχή την ανθρωπιστική βοήθεια και συνεχίσουμε τη δουλειά που έχει ξεκινήσει η Ιταλική Προεδρία για την ενίσχυση συνεργασία μεταξύ ανθρωπιστική βοήθεια και αρχών, αρχών ανθρωπιστική βοήθεια και αρχών πολιτική προστασία. Κάτι το οποίο μπορεί να ε, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση τη αντοχή αυτή τη βοήθεια και τη δράση σε χώρε που κινδυνεύουν προ τώρα από κρίσει. Ιδιαίτερα για τη διαχείριση των φυσικών ε, καταστροφών έχουμε εστιάσει τους ε, στόχους μας για την παγκόσμια διάσκεψη για τον περιορισμό των φυσικών καταστροφών DRR που πρόκειται να γίνει το Μάρτιο στην Ιαπωνία. Παρακολουθούμε δε ως Προεδρία ιδιαίτερα προσεκτικά την προετοιμασία της διάσκεψης και σκοπεύουμε μαζί με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουμε το follow-up. Η τέταρτη προτεραιότητά μας είναι να συνεισφέρουμε στις προετοιμασίες ε, ε, της ανθρωπιστική ανθρωπιστικής Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη τον επόμενο χρόνο. Ε, έχει, είναι μοναδική ευκαιρία για να βρούμε ποιοι είναι οι τρόποι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ουγγρική και η Φιλανδική κυβέρνηση ε, θα φιλοξενήσουν την Περιφερειακή Σύνοδο Διαβούλευσης Ευρώπης και άλλων, της Ομάδας Ευρώπης και άλλων στο Βουδαπέστη 3 και 4 Φεβρουαρίου, ενώ η Γερμανία θα φιλοξενήσει ένα θεματικό, μια θεματική συνεδρίαση διαβούλευση το Σεπτέμβριο. Ε, εμείς ως Προεδρία θα διασφαλίσουμε ότι οι συζητήσεις στην ε, Βουδαπέστη θα τύχουν τις κατάλληλες παρακολούθησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ανοίξουν το δρόμο για άλλε προετοιμασίε για την ε, Σύνοδο κατά τη διάρκεια των επόμενων Προεδριών Λουξεμβούργου και Ολλανδίας. Επίσης να πω και για το θέμα της ε, πρωτοβουλίας ε, των εθελοντών ενίσχυση βοήθεια τη Ευρωπαϊκής Ένωση, που ξέρω ότι σας την υποστηρίξατε με ενθουσιασμό. Χαίρομαι ε, που οι προτάσεις της Κομισιόν για εφαρμοστικές ε, πράξεις και πράξεις αντοξιοδότηση έγιναν δεκτές. Ε, αυτή η πρωτοβουλία παίρνει ορμή και όθηση και θα φτάσουμε πολύ σύντομα σε απτά αποτελέσματα. Ε, θα περιμένουμε να λάβει χώρα η πρώτη να δημιουργηθεί η πρώτη ομάδα εθελοντών παρόλο που δεν θα γίνει υπό τη δική μας προεδρία. Ε, η περίοδος αυτή είναι περίοδος μεγάλων προκλήσεων αλλά και ευκαιριών. Ε, έχουμε πολλές ε, κρίσεις, ανθρωπιστικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα είναι και ευκαιρία διότι πλησιάζουμε στην Σύνοδο Κορυφής του 2016, την Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής, και εμείς θα εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει το ρόλο της για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να υποφεληθεί από τις ευκαιρίες. Γνωρίζω ότι... Α, σχολίασα μόνο ορισμένα από τα πιο σημαντικά θέματα, οπότε περιμένω τις δικές σας ερωτήσεις και παρατηρήσεις για αυτά ή για άλλα ανθρωπιστικά ζητήματα. Περιμένω τους επόμενους έξι μήνες να συνεργαστούμε στενά και περιμένω επίσης και να γίνει μια πολύ ευχάριστη συζήτηση και ωφέλιμη συζήτηση τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επισκόπηση. του προγραμματός σας για το επόμενο εξάμεινο. Δύο μιλτές. Καταρχήν ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ και την ε, Υπουργό. τόσο για την ε, Προεδρία όσο και για τις δικές προσωπικές προσπάθειες να είναι σε επαφή μαζί μας. μας παρουσίασε τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας. Αναφέρατε μεταξύ άλλων κρίσεων και την Ουκρανία. Θα ήθελα να σας στηρίξουμε και να στηρίξουμε και τις προθέσεις του Επιτρόπου Στυλιανίδη ε, που έχει σκοπό να επισκεφθεί την Ουκρανία. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο από το Κοινοβούλιο. Επίσης, αναφέρατε τις χώρες που έχουν πληγεί από τον έμπολα. Έχουν από δύο πράγματα. Χρειάζεται συνεχή στήριξη, διότι θα πρέπει να αποφύγουμε να ξεχάσουμε το πρόβλημα επειδή δεν είναι τόσο επίγον και απειλητικό πια. Και το δεύτερο είναι ότι η Κομισιόν στις πρώτες φάσεις της κρίσης ε, δήλωνε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξύνεται αλλά τα κράτη-μέλη είχαν καθυστερήσει να απαντήσουν και να ανταποκριθούν. Και ο διορισμό του κ. Στυλιανίδη ω συντονιστή ήταν πολύ καλό βήμα. Αλλά πώ θα συνεχιστεί στο μέλλον αυτό ο συντονισμό. Τέλο. Διαθέτουμε πλέον τον προπολογισμό για τον τρέχοντα χρόνο. Αλλά ποια είναι η επιθυμία των κρατών μελών έτσι ώστε να μειωθεί η διαφορά ανάμεσα στα ποσά τα οποία έχουν υποσχεθεί για δωρεές και αυτά τα οποία εκταμείευονται πραγματικά. Ευχαριστώ. Okay, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ. Καταστήσατε σαφές ότι προσφέρετε συνεργασία, κάνετε πρόταση για συνεργασία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο το είδαμε αυτό ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πολύ για το ότι ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου δραστηριοποιήσετε τόσο γρήγορα για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στην μονιμότητα της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση βέβαια στον προϋπολογισμό, αλλά κάθε φορά πρέπει να ε, κάνουμε μεγάλο αγώνα για να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Εάν δούμε πόσο αδύρυτες είναι οι ανάγκες σε διάφορες περιοχές του κόσμου, τα Ηνωμένα Έθνη ξέρουμε ότι είναι ούτως ή άλλως ε, σε κατάσταση υποχρηματοδότησης, η κατάσταση στους καταβλισμούς των προσφύγων είναι φρικτή, βλέπουμε ότι χρειάζεται να καλύψουμε πολύ χαμένο έδαφος. Ε, είχαμε πριν από εσά τον κύριο Σόλχαϊμ από τον ΟΣΑ εδώ και ο οποίος μας είπε ότι έχουν σημειωθεί πολλές πρόοδοι σε πολλούς τομείς, αλλά όχι στη χρηματοδότηση και ιδιαίτερα σε πολλά κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι υπάρχει έως και οπισθοδρόμηση στη χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ιδιαίτερα θέλω να αφαιρθώ βέβαια στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ε, πάντοτε επικρίνεται για την επιφυλακτική έναντι της Ευρώπης θέση του. Αλλά στον τομέα τη ανθρωπιστικής βοήθειας ο Κάμερον και το Ηνωμένο Βασίλειο νομίζω ότι μπορούν να χαρακτηριστούν ω υπόδειγμα. Ε, Εμεί στη Γερμανία με διαφορετικέ τα τελευταία 15 χρόνια κυβερνήσει δεν μπορέσαμε να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον στόχο του 0,7% ούτε με φιλελεύθερη ούτε με σοσιαλδημοκρατική ε, η σοσιαλδημοκρατική μαζί με φιλελεύθερη ή με σοσιαλδημοκρατική μαζί με τη χριστιανοδημοκρατική ή με σοσιαλδημοκρατική μαζί με πράσινη ε, με πράσινο κόμμα κυβέρνηση δεν μπορέσαμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας στην αναπτυξιακή βοήθεια στην, ε, τελευταία ανάλυση αξιοπιστία μας ως προς την στράτευσή μας αυτή. Για δε τα ανθρωπιστικά σχέδια και έργα σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν πολλές αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταλανίζονται ε, από τους περιορισμούς τους οικονομικούς. Χρειάζεται να ε, αναβάλουν την εκτέλεση πολλών έργων τους. Αυτό βέβαια θα υποφέρει και η αξιοπιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές είναι αντιπροσωπείες οι οποίες ε, αναγκάζονται να μην καταβάλουν τα ποσά που έχουν δεσμεύσει για τα οποία έχουν δεσμευστεί μάλλον και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό ήθελα να το αναφέρω. και εν ώψη της ε, προβλεπόμενης ε, συνεδρίασης ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όμως αναβλήθηκε γιατί δεν θέλησαν ορισμένα κράτη-μέλη να ε, διεξαγάγουν σε στη διάρκεια μιας προεδρίας τους, Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και έτσι τώρα έχουμε δύο συνεχιζόμενες συνόδους ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτος ΑΚΕ. Ελπίζω εσείς να θέσετε στο επίκεντρο του θεματολογίου σας και το θέμα της ΑΚΕ και να δούμε με τη Λεπτονική Προεδρία μια εικόνα διαφορετική από αυτή που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Και έτσι κάτι άλλο, πολύ σημαντικό που αναφέρατε, την πρωτοβουλία για τους εθελοντές στην Ευρώπη. Πολύ ενδιαφέρον, αν την υποστηρίζετε, αλλά συγκεκριμένα η Λετωνία τι κάνει για να ενισχύσει αυτό το σώμα των εθελοντών. Θα ακούσουμε μία ακόμα ερώτηση σε αυτό το γύρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ την Υπουργό από τη Λετωνία. Καλή τύχη σας εύχομαι για το εξάμεινο της Λετωνικής Προεδρίας. Ήδη είχαμε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε και στο Στρασβούργο και είδαμε πραγματικά ότι έχετε όρεξη για δουλειά, για εργασία. Να αναφερθώ τώρα σε ένα σημείο. Ξεκινάω βέβαια από την γενικότερη πολιτική βούληση που υπάρχει συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ζητήματα ανάπτυξης. Θα ήθελα όμως πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ζητήματα της ανάπτυξης, για την έννοια της ανάπτυξης. Όπως είπε ο κύριος ε, Νόιζερ, Νομίζω ότι η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ μικρή για κάποια προγράμματα, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο πώς εμείς προσεγγίζουμε την ανάπτυξη αυτή καθ' αυτή, αλλά πώς υλοποιείται τελικά η ανάπτυξη. Γιατί αν τελικά χρηματοδοτούμε τόσο λίγο μία πολιτική η οποία βασίζεται τελικά και στην χρηματοδότηση, μάλλον και στον προπολογισμό που έχουν τα κράτη-μέλη, τα, μάλλον τα, μέλη, τα κράτη εκείνα τα οποία α, λαμβάνουν την βοήθεια αυτή, θεωρώ ότι η δική μας η μικρή συμβολή είναι κάπως υποκριτική. Αντίθετα, νομίζω ότι στα πλαίσια της ατζέντα ανάπτυξης θα πρέπει να υπάρχει και μία κάποια επικοινωνία, μία ενημέρωση όσον αφορά τη λεγόμενη υπεύθυνη κατανάλωση. Δηλαδή, θα πρέπει ορισμένες χώρες, ιδίως οι χώρες οι οποίες λαμβάνουν τη χρηματοδότηση από εμά να συνειδητοποιήσουν ότι με συγκεκριμένα μοντέλα οικονομία και κατανάλωση δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν κοινωνίε ευημερία. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάμε περισσότερο και για το ζήτημα αυτό, το οποίο θεωρώ ότι είναι θεμελιώδε και συνδέεται άμεσα με την ίδια την έννοια τη ανάπτυξη. Μπορούμε να ακούσουμε απαντήσει για τι τρει αυτέ ερωτήσει. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να απαντήσετε αν θέλετε και εσείς πρώτα σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις και μετά να κάνουμε ένα επόμενο γύρο ερωτήσεων. So, uh, thank you for, for, uh, Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω καταρχάς στην ε, ερώτηση του κυρίου Στίερ. Αναφερθήκατε στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια στον ιό του έμπολα. Ξέρετε ότι ήδη την ε, προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ε, ανταπόκριση στην ανθρωπιστική κρίση που έχουμε στην Ουκρανία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε και ένα ψήφισμα Όσον αφορά συγκεκριμένα λοιπόν ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία, αυτό προφανώς θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Λετωνική Προεδρία. Πέρυσι, το σύνολο της αρρωγής προς την Ουκρανία ήταν περίπου 76 και πάνω μάλλον από 76 εκατομμύρια ευρώ και τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να δίνουν αρρωγή προς τη χώρα αυτή και να αντιμετωπιστούν βασικές ανάγκες βασικές ανάγκες του πληθυσμού, ιδίως στις περιοχές εκείνες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση, από την ένοπλη σύραξη και ήδη από πέρυσι είχαμε δεσμευθεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα δίναμε συγκεκριμένα προϊόντα, θα παρήχαμε συγκεκριμένα αγαθά προς τους πολίτες της χώρας αυτής. Ενισχύουμε πάντως την ανθρωπιστική μας εργασία και συντονίζουμε τη δράση μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου υπάρχει συντονισμένη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη και θέλουμε να ενισχύσουμε περισσότερο και την προβολή της ανθρωπιστικής βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Τώρα όσον αφορά τον ιό εμπόλα, Προφανώς και αυτός αποτελεί προτεραιότητα του Συμβουλίου. Θα συνεργαστώ επίσης με τον αρμόδιο επίτροπο. Ήδη την έχω συναντήσει και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια στενή συνεργασία. Η εμφάνιση του ιού αυτού στην Δυτική Αφρική εξελίχθηκε τελικά σε ευρύ ανθρωπιστική κρίση που επηρεάζει πολλές οικονομίες και πολλά κοινωνικά συστήματα σε όλες τις χώρες που έχουν πληγεί στην ευρύτερη εκείνη περιοχή. Χαιρόμαστε που υπάρχει μια ενεργή όμω συμμετοχή των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του ιού αυτού και ήδη βλέπουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Πρόσφατα το Μάλι κηρύχθηκε ως χώρα απαλλαγμένη από τον ιό έμπολα, αφού βέβαια είχε πληγεί τουλάχιστον για μια περίοδο 42 ημερών από τον ιό αυτό. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε την επέκταση του ιού αυτού και θα πρέπει στη συνέχεια να υποστηρίξουμε την ε, μακροπρόθεσμη ανάκαψη των χωρών που έχουν πληγεί από τον ιό αυτό. Βασικό στόχο λοιπόν τη δική μα Προεδρία θα είναι να δούμε ποιε είναι οι μακροπρόθεσμε επιπτώσει του ιού αυτού, τη επιδημία αυτή στι χώρε τη Δυτική Αφρική και πώ επηρεάζει τα κοινωνικά και τα οικονομικά συστήματα των χωρών αυτών. Θα προσπαθήσουμε επίσης να αντλήσουμε και τα απαραίτητα διδάγματα από την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Και βέβαια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε και από την διεθνή ανταπόκριση στον ιό έμπολα. Ακούστηκαν διάφορες επικρίσεις για τη δράση των ε, Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και για την ε, έλλειψη συντονισμού που υπήρξε στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν στην επόμενη συζήτηση που θα γίνει μεταξύ Ηνωμένων Εθνών αλλά και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας προκειμένου να μην επαναληφθούν τα λάθη αυτά στο μέλλον. Τώρα έρχομαι στις ερωτήσεις του κυρίου, του κυρίου Νόιζερ όσον αφορά την έλλειψη χρηματοδότησης και όσον αφορά το ζήτημα της ε, συνέλευσης, ε, της κοινωνικής συνέλευσης εκπροσώπησης και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα αναφερθώ επίσης και στο ζήτημα της υποστήριξης των προσφύγων από τη Συρία. Και θα αναφερθώ επίσης και στα ερωτήματά σας όσον αφορά τα προγράμματα επισητιστικής βοήθειας στη Συρία. Αναφερθήκατε επίσης στον προπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρώτον λοιπόν, όταν αφαιρόμαστε στους πρόσφυγες ε, από τη Συρία προφανώς θέλουμε να υποστηρίξουμε τα εκατομμύρια των προσφύγων που έχουν ε, φύγει, έχουν πάει σε γειτονικέ χώρες. Γνωρίζουμε ότι η Ορδανία, ο Λίβανος, η Τουρκία και οι άλλες όμερες χώρες θα πρέπει να υποστηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τις επιτόπου ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας. Πέρυσι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ε, ανησυχήσει από την ε, εξαιτία της ε, προσωρινής αναστολής των προγραμμάτων επιστηστικής βοήθειας προς τους Σύριους πρόσφυγες. Το καλό είναι ότι τα προγράμματα αυτά άρχισαν πλέον πάλι να λειτουργούν και αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και κατά αυτόν τον τρόπο καλύψαμε το κενό το οποίο είχε προκύψει στην χρηματοδότηση των επισητιστικών προγραμμάτων για τους πρόσφυγες. Όσον αφορά τώρα τον ευρύτερο προπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό 2015 ολοκληρώθηκαν και ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία όσον αφορά τον προπολογισμό. Χαιρόμαστε επίσης που υπάρχει μια συμφωνία και τον, για τον διορθωτικό προπολογισμό του 2014 και έχουμε επιπλέον 250 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Στα πλαίσια του προπολογισμού 2015 προβλέπονται αντίστοιχα ποσά όσον αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων και τις πληρωμές για την ανθρωπιστική βοήθεια και κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα αποφύγουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια του 2014. Η Προεδρία επίσης ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση προκειμένου να υποστηρίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και το, τα καλεί επίσης να ανταποκριθούν στην υποχρέωση του 0,7% από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους, το οποίο θα πρέπει να δίδεται με τη μορφή ODA, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Ξέρετε ότι η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας εξαρτάται πάρα πολύ από αυτή την εθνική συνεισφορά και μάλιστα τον Ιούλιο θα έχουμε και μία σύνοδο με το ζήτημα αυτό ακριβώς, τη χρηματοδότηση δηλαδή της αναπτυξιακής βοήθειας. Η Προεδρία λοιπόν θέλει να συμβάλλει προκειμένου να προετοιμάσει την διεθνή αυτή σύνοδο Financing for Development και θα έχουμε και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο όπου θα γίνει μια πολιτική συζήτηση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος που θα πρέπει να δίδεται από τα κράτη-μέλη με τη μορφή επίσημης αντιξιακής βοήθειας. Εφόσον κάνουμε εμείς αυτή τη ζήτηση το Μάρτιο θα είμαστε και πιο προετοιμασμένοι για τη σύνοδο του Ιουλίου. Αναφερθήκατε επίσης στην συμβολή της λετονικής Προεδρίας όσον αφορά την εθελοντική ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλουμε και εμείς να προωθήσουμε την εθελοντική εργασία και να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχει, υπάρχουν, με συγχωρείτε, προκειμένου να βοηθήσουμε πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ανθρωπιστικές δράσεις να το πράξουν. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις του κυρίου Νόιζερ. Α, ναι, ΑΚΕ. Όσον αφορά πάλι την ε, ανθρωπιστική βοήθεια, προφανώς δεν λησμονούμε τις χώρες ΑΚΕ και ενθαρρύνουμε πάλι τα κράτη-μέλη να διοργανώσουν τις επόμενες συνεδριάσεις ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Επί του παρόντος προσπαθούμε να δούμε ποιος θα εκπροσωπήσει τη δική μας την Προεδρία στην επικείμενη συνεδρίαση. Δεν έχουμε πάρει κάποια σχετική απόφαση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο Υπουργός Εξωτερικών της Λετωνίας θα συμμετάσχει ο ίδιος στη σύνοδο αυτή. Ας περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις του κυρίου Κοράου. Καταρχάς, όσον αφορά την παρατήρησή σας για την επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, εντελώ ε, ευχάριστα βρίσκομαι εδώ πέρα και συνεργάζομαι μαζί σας και εγώ όντας πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ε, Λετωνικού Κοινοβουλίου συμμετείχα ιδιαίτερα σε συζητήσεις που είχαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να συνεργάζομαι και να μιλώ ανοιχτά με του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την χρηματοδότηση τη ανθρωπιστική βοήθεια, νομίζω ότι η ερώτησή σα σχετίζεται με την ερώτηση που έθεσε ο κύριο Νόιζερ για τον προπολογισμό τη ανθρωπιστική ανάπτυξη, όπω σα είπα θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι για τη διεθνή διάσκεψη Financing for Development που θα λάβει χώρα τον Ιούλιο προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε όλο και πιο αποτελεσματικά να χρηματοδοτούμε τις διάφορες δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Όσον αφορά τώρα την Παγκόσμια Σύνοδο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, είπα στις αρχικές μου παρατηρήσεις ότι όντως υπάρχουν κάποιες αδυναμίες το Παγκόσμιο Σύστημα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και επομένως στη Σύνοδο του 2016 θα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία για να δούμε πώς μπορούμε παγκοσμίω να βελτιώσουμε το σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας. Στη Σύνοδο αυτή θα συμμετέχουν δωρητές, χώρες δικαιούχοι, αλλά και άλλοι εταίροι, ακαδημαϊκοί καθηγητές, μη εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στα πλαίσια λοιπόν του Συμβουλίου θα διεξάγουμε συζητήσεις οι οποίες ήδη ξεκίνησαν και κατά τη διάρκεια του 2014 με τις προηγούμενες προεδρίες και ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες συνεδριάσεις ε, διαβουλεύσεων για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε όλο και καλύτερα προετοιμασμένοι σε αυτή τη σύνοδο. Έχουμε τέσσερις ακόμα μιλητές, πέντε, για να έχουμε την κυρία Χόιμπερκ, Βάρινεν, Ζαμπόφσκα, και άλλους δύο μιλητές, πέντε. Δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος. Μαρία Χόιμπρουκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις. Όταν μιλούμε για μια διαρκή υποχρηματοδότηση Καλό είναι βέβαια να λέτε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή μαζί, να συνενωθούν οι προσπάθειες, έχετε κάνει την ανάλυση, έχετε μιλήσει για την αξιολόγηση των αναγκών. Υπάρχει όμως κάποιο σχέδιο για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό και στην πράξη, πώς μπορεί να υλοποιηθεί στα διάφορα κράτη. Γιατί το θέμα σε σχέση με τον έμπολα είναι να κοιτάξουμε και βέβαια πώς θα αντιμετωπίσουμε την επέκταση της επιδημίας, αλλά θα έπρεπε και προκαταβολικά να κάνουμε τη σχετική επένδυση. Ερωτώ λοιπόν για αυτό και επίσης για το σώμα των εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας. Πώς θα λειτουργήσει, προβλέπετε κάποιο τύπου συντονισμός, γιατί και στην περίπτωση του έμπολα υπήρχε υποτίθεται συντονισμό, αλλά σε αυτό ακριβώ ειστερούσαμε, ότι δεν υπήρξε επαρκή συντονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Βαρινέν, ε, θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για τις α, ανθρωπιστικές ανάγκες που δημιούργησε η κρίση στην Ουκρανία. Φαντάζομαι ότι στον Τόνπας είναι επικρατεί η πιο δύσκολη κατάσταση. Ε, βέβαια έχουμε ανθρώπους που έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους σε πολλά άλλα σημεία της Ουκρανίας και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Ρωσία. Ποια είναι η κατάσταση γενικά ε, των διαφόρων ομάδων ε, του πληθυσμού που έχουν πληγεί και ποιες, ποια είναι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους βοηθήσει. Κυρία Αναζεμπόφσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Λουκατσέβισκα. Θα ήθελα να σχολιάσω την τρίτη προτεραιότητα που αναφέρατε. την ε, σχέση ανάμεσα στην ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά τα δύο συνδέονται πολύ στενά και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν πρέπει να χωρίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες ζουν 4,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. 2 δισεκατομμύρια μεταξύ αυτών ε, είναι ασθενείς με φυματίωση. 600 εκατομμύρια πλήττονται, ομολύονται από ελονοσία κάθε χρόνο. 50 εκατομμύρια με Και 10 εκατομμύρια το χρόνο μεταξύ αυτών πεθαίνουν από πείνα. Κοιτάζοντας αυτά τα στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι πέραν των θεομηνιών που οδηγούν σε ε, ανθρωπιστικές κρίσεις. Η φτώχεια και τα προβλήματα υγείας είναι ε, οι άλλοι δύο λόγοι που δημιουργούν ανθρωπιστικές κρίσεις. Ο έμπολα ε, δεν ε, ε, αναπτύχθηκε τόσο πολύ σε άλλες χώρες, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα σε αυτές, για συγκεκριμένους λόγους. Αυτές οι χώρες, ε, οι οικογένειες προς αυτές τις χώρες ζουν σε συνεχή αγωνία. Ε, δεν ξέρουν καν τι, θα, τι, τι φαΐ θα δώσουν την επόμενη μέρα στα παιδιά τους και μάλιστα αυτό τους οδηγεί και μια σε μια σχετική απάθεια διότι είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται. Συνεπώς θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα μιλήσετε και για την ε, ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα την ε, εκπαίδευση και την επιμόρφωση των γιατρών, των νοσοκόμων, του ιατρικού προσωπικού γενικότερα. Σίγουρα η ανάπτυξη αυτή τη εκπαίδευση θα πρέπει να είναι μόνιμη προσπάθεια, αλλά κάθε Προεδρία πιστεύω θα πρέπει να κάνει τη δική της προσπάθεια να επενδύσει ε, χρήματα για την ε, βελτίωση του τομέα της υγείας. Γιατί δάλλος ε, δεν πρόκειται ποτέ αυτές οι χώρες να βγουν από τον φαύλο κύκλο ε, που τις μαστίζει εδώ και δεκαετίες. Ευχαριστώ. να ακούσουμε άλλε δύο ερωτήσεις και τα σχόλια, τις απαντήσεις μετά. Τέλει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχόμαι καλή επιτυχία στη Λετωνική Προεδρία σας σημαντικό το έτος και μεγάλες προκλήσεις. Είπατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος ε, για την ανάπτυξη φέτος ξεκίνησε στη Ρήγα. Το Ευρωπαϊκό Έτος για την ανάπτυξη όμως δεν θα πρέπει να είναι μόνο μια ευκαιρία ορισμένοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ή όργανα να ασχοληθούν με την αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση, μια δημόσια εκδήλωση για να διεκδικήσουμε περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια σε περισσότερους τομείς το, της πολιτικής ζωής στην Ευρώπη. Το multi-level governance δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές και φορείς πρέπει να εγγραφούν σε αυτόν τον αγώνα. Ξέραμε βεβαίως ότι το 2015 θα είναι το έτος της ε, αναπτυξιακής ε, βοήθειας από καιρό. Ωστόσο το θέμα είναι σχετικά γνωστό στο ευρύ κοινό. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν και πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε ώστε και οι, ε, οι ομότιμοι σας, οι ομολογοί σας στο Συμβούλιο να ενδιαφερθούν περισσότερο, να κοινοποιήσουν, να καταστήσουν πιο γνωστό τον αγώνα αυτόν για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ευρώπη και επίσης φέτος θα έχουμε και τις διαπραγματεύσεις για την ε, Διατλαντική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και Επενδύσεων, την TTIP. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες εκφραζόμενες από τα αναπτυσσόμενα κράτη που φοβούνται ότι θα μείνουν εκτός παιδείας. Ε, ίσως λοιπόν θα έπρεπε εδώ να μην παραμελήσουμε τις επαφές με τους εταίρους μας στα αναπτυσσόμενα αυτά κράτη ώστε να τους ε, διαβεβαιώσουμε πως στο μέλλον, εάν υλοποιηθεί βέβαια αυτή η συμφωνία, δεν θα έχει δυσμενείς συνέπειες στη δική τους εμπορική θέση έναντι της Ευρώπης, ότι, θα, ότι δεν θα δυσχερανθεί δηλαδή η πρόσβασή τους σε αγορές σε σχέση με αυτό που έχουν τώρα. Η αναπτυξιακή βοήθεια είναι πολύ σημαντική βεβαίω, αλλά χρειάζεται και πρόσβαση στι αγορέ τη Ευρώπη για τα κράτη αυτά. Δεν μπορεί δηλαδή να εξαντλείται η αναπτυξιακή πολιτική στην ε, απλή διοχέτευση κάποιων ε, πλεονασμάτων στην παραγωγή τη γεωργική των ΗΠΑ προς τους ε, λιμοκτονούντες πληθυσμού των φτωχών κρατών. Τα τελευταία χρόνια συζητούμε συνέχεια το αν θα ξανά συναυθεί μια νέα συμφωνία κοτονού ή αν θα ξανά ε, γίνει διαπραγμάτευση από το μηδέν. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και στη διάρκεια αυτή τη θητεία ιδιαίτερα να δώσουμε ιδιαίτερη έφαση στα μεγάλα στου μεγάλους στόχους. Είναι μικρό κράτο η Λετωνία και το ξέρω. Ξέρω ότι σε σχέση με τα μεγαλύτερα κράτη έχει σωσπεριορισμένο περιορισμένο διοικητικό δυναμικό, διαχειριστικό δυναμικό, αλλά έχει τεράστια ικανότητα πολιτική, ηθική, αλλά και ε, πνευματική ώστε να έρθει αντιμέτωπη και να κερδίσει τον αγώνα σε, αυτά, σε αυτούς τους μεγάλους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φουνσουλίκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ την ε, Υπουργό για την παρουσίασή της. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τη στρατηγική προσέγγιση της Λετωνικής Προεδρίας προς την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί δεν ήταν πολύ σοφές Για μένα το ποια είναι τα κύρια, ποια είναι, τα κύρια θέματα, οι κύριοι τομείς που έχετε ορίσει στις προτεραιότητές σας. Λέτε ότι Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά ξέροντα ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι που έχουμε στη θέση μα για την ανθρωπιστική βοήθεια στην προσεχή δημοσιονομική περίοδο, μπορείτε να δώσετε απαντήσεις με συγκεκριμένη εστίαση στις κύριες προτεραιότητες της Λεωτονικής Προεδρίας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Κύριε Υπουργέ, ακούσατε πολλές ερωτήσεις. Σας ακούμε λοιπόν για τις απαντήσεις σας. Όντως πολλές ερωτήσεις λέει η Πρόεδρος. Ελπίζουμε να καταφέρετε να απαντήσετε σε όλες. Με την κυρία Χόιμπροκ ξεκινάμε και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πολύ. όσον αφορά τις ερωτήσεις της κυρίας Χόιμποκ. Για μια σφαιρική προσέγγιση. Η Προεδρία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των εξωτερικών κρίσεων και διενέξεων. Υπάρχει ένα σχετικό σχέδιο δράσης το οποίο θα αναπτύξει η ύπατη εκπρόσωπος μέσα, στα, μέσα στο 2015, το τρίτο τρίμηνο του 2015, Πρέπει όμως να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι αποτελεί εξωτερική πολιτική και τι αποτελεί ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπου, δηλαδή να είναι ξεχωριστές οι δράσεις αυτές. Όσον αφορά τώρα το σώμα των εθελοντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα υποστηρίξουμε την εθελοντική αυτή εργασία στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των υφιστάμενων δομών. Δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία σύγχυση και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός όλων των εταίρων χωρίς επικαλύψεις, χωρίς να περιπλέκουμε τα πράγματα. Τώρα, η διασύνδεση ανάμεσα σε ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας και και αναπτυξιακής βοήθειας. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και τις δύο πτυχές στα πλαίσια της σφαιρικής προσέγγισης και νομίζω ότι υπήρξε και άλλη μία ερώτηση όσον αφορά τη διασύνδεση ανάμεσα στα ζητήματα ανάπτυξης και τα ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Το ζήτησα, μάλλον το συζήτησα αυτό και με τον Επίτροπο Μίμικα και με τον Επίτροπο Στυλιανίδη, τους δύο αρμόδιους δηλαδή επιτρόπους για τις δύο αυτές πολιτικές και είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολύ θετική συνεργασία ανάμεσα στους δύο αυτούς τομείς. Ανθρωπιστική βοήθεια από τη μια, αναπτυξιακή βοήθεια από την άλλη. Όχι μόνο για κάποιες άμεσες βραχυπρόθεσμες δράσεις, αλλά και για την εξέβρεση μακροπρόθεσμων λύσεων και για την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τον ιό έμπολα, προσπαθούμε προφανώς στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας να καλύψουμε τις άμεσες συνέπειες, να θεραπεύσουμε τις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις, αλλά στα πλαίσια της ανεπτυξιακής βοήθειας στη συνέχεια μπορούμε να προβούμε σε κάποιες πιο μακροπρόθεσμες δράσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με ζητήματα όπως ε, η υγιεινή, το σύστημα υγείας, το σύστημα αποχέτευσης ορισμένων πόλεων. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι δράσεις μπορεί να βοηθήσουν όντως συγκεκριμένε χώρες να αναπτύξουν την υποδομή την οποία θα χρειαστούν ούτως ή άλλως για το μέλλον τους. Όχι μόνο στα πλαίσια της αντιμετώπισης μιας κρίσης. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Βαρίνεν, ελπίζω ότι ε, προφέρω σωστά το όνομά σας. Μιλήσατε για την Ουκρανία, καθώς επίσης και για τις ανάγκες του Ουκρανικού λαού. Προφανώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει έρθει πια ο χειμώνας και ότι ο Ουκρανικός λαός δεν έχει μόνο ανάγκες που έχουν να κάνουν πλέον με την υγειονομική περιθέρψη, αλλά πρέπει να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν και τον δρυμή χειμώνα, που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα για τους ανθρώπους όπως το καταλαβαίνετε. Όπως είπα λοιπόν και στην παρέμβασή μου, η κυβέρνηση της Λετωνίας ήδη έχει παράσχει χρηματοδότηση και ενθαρρύνει και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχουν αντίστοιχη χρηματοδοτική βοήθεια και εμείς ως Προεδρία στη συνέχεια θα θέλαμε να συντονίσουμε την συμβολή αυτή από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα τώρα προκύπτει ακόμα πιο έντονο στις περιοχές εκείνες που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση, καθότι για παράδειγμα δεν καταβάλλονται συντάξεις στις ε, περιοχές αυτές οι οποίες δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, έχουν προκύψει και πολλά άλλα προβλήματα για τον Ουκρανικό λαό που ζει σε αυτές τις περιοχές και που ουσιαστικά βλέπει τα εισοδήματά του να μειώνονται συνεχώς. Στο Συμβούλιο λοιπόν Ευρωπαϊκών, ναι, συγγνώμη, Εξωτερικών Υποθέσεων την Δευτέρα προσπαθήσαμε να δούμε τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το πρόβλημα. Προφανώς θα πρέπει να βρούμε λύσεις για την Ουκρανία αυτή καθ' αυτή, συνολικές δηλαδή λύσεις, αλλά και πιο συγκεκριμένε λύσεις όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον Ουκρανικό λαό. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση των προσφύγων, πάλι τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και σίγουρα δεν είναι εύκολα και βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα. Σίγουρα η κατάσταση είναι αρκετά σαφής, πολύ πλοκή και είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να βοηθήσει την Ουκρανία για να επιλύσει την κατάσταση που έχει προκύψει και στις σχέσεις με τη Ρωσία αλλά και για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή προκειμένου να καταφέρει να αναπτυχθεί και να επιληθεί η ανθρωπιστική κρίση που έχει προκύψει κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Αναφέρομαι τώρα σε ερωτήσεις κυρία Ζαμπόρσκα. Κυρία Ζαμπόρσκα, αναφερθήκατε και εσείς στον ιό του έμπολα. Νομίζω ότι έδωσα επαρκείς απαντήσεις. Επαναλαμβάνω ότι όντως θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Δυτική Αφρική αλλά και σε άλλες περιοχές και σε αυτό θα επικεντρωθούμε στη διάσκεψη θα λάβει χώρα στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και χρηματοδότηση αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες αυτές. Τώρα, όταν αναφέρθηκα στο έτος ανάπτυξης, κύριε Τσέλερ, εσείς αναφερθήκατε στο έτος αυτό, ξέρετε ότι συζητήσαμε το ζήτημα και στην προηγούμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ακούσαμε και την κυρία Μογκερίνη, την τη εκπρόσωπο, η οποία αναφέρθηκε στο ζήτημα της αναπτυξιακής βοήθειας και όπως είπε και η πρόεδρό σας, στις 9 Ιανουαρίου κηρύξαμε επίσημα την έναρξη του έτους ανάπτυξης, ένας από τους βασικούς στόχους του έτους αυτού είναι να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες για ζητήματα ανεπτυξιακής βοήθειας. Στόχος μας είναι να εμπλέξουμε όλο και περισσότερο τους φορείς της κοινωνίας, την τοπική κυβέρνηση, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις από διάφορα κράτη-μέλη προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι πολίτες, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς κύριε Τσέλερ. και θα προσπαθήσουμε βέβαια να διαφημίσουμε και να προβάλλουμε και να προωθήσουμε το έτος αυτό και στη Λετωνία αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε μεμονωμένα κράτη-μέλη τα οποία ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υποβάλλουν σχέδια ανάληψης δράσης στα πλαίσια του έτους αυτού. Και υπάρχουν από ό,τι βλέπω όλο και περισσότερα κράτη-μέλη τα οποία θα εγκαινιάσουν κάποια νέα σχέδια δράσης για το σημαντικό αυτό έτος ανάπτυξης. Πάλι η πρωτοβουλία αυτή όμως προέκυψε από τον τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις λετονικές μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις καθώς επίσης και τη λετονική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που βοήθησε και αυτή με τη σειρά της να προωθηθεί το έτος ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, περαιτέρω βοήθεια και συνεισφορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να προβάλλουμε ευρύτερα το έτος αυτό ανάπτυξης. Και κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα προσελκύσουμε και περισσότερους φορείς και περισσότερους πολίτες να ενεργοποιηθούν στα ζητήματα αυτά τα οποία υπάγονται στο έτος ανάπτυξης. Αναφερθήκατε επίσης στο ζήτημα του εμπορίου. Το ζήτημα αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο, είναι αρκετά επίκαιρο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το εξαντλήσουμε ή να τον άλλο στη σημερινή συνεδρίαση να καλύψουμε πλήρως το ζήτημα αυτό. Περνάμε αν θέλετε και σε τομείς διαφορετικής πολιτικής αυτή την φορά. Πάντως στα πλαίσια της Επιτροπής Ίντε θα είμαι σε θέση με εσά και με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας να μιλήσω περισσότερο για ζητήματα εμπορίου. Πάντως, το εμπόριο είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το εμπόριο προωθεί προφανώς την οικονομική ανάπτυξη, προωθεί την οικονομική μεγέθυνση. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ισότιμοι όροι εμπορίου υφίστανται και ότι θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να υποφεληθούμε από τον θεμητό ανταγωνισμό και από τις ε, θεμητές αυτές ε, εμπορικές συναλλαγές ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ως χορηγή των ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Περνάω τώρα στα τελευταία ερωτήματα. το οποίο είπε ο κύριος Φρουντσουλίτσα. Ελπίζω πάλι να προφέρω σωστά το όνομά σας όσον αφορά τις προτεραιότητες της ελετονικής Προεδρίας. Ξέρετε ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενός αξιωματούχου τουλάχιστον, είναι να προφέρει σωστά τα ονόματα των ε, άλλων αξιωματούχων. Φραντζούλικα λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με βοηθήσετε να προφέρω σωστά το όνομά σας. Λοιπόν, οι προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας. Προφανώς θέλουμε να ανταποκριθούμε στις διάφορες κρίσεις. Έχουμε πολύ σημαντικές σοβαρές κρίσεις. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε έναν αποτελεσματικό συντονισμό και να αποφύγουμε να προκύπτουν κενά και χάσματα στην ανταπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι προφανώς σημαντικότερη προτεραιότητα για μας. Θέλουμε επίσης να τηρήσουμε τις αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας, το ζήτημα της πρόθεσης της ανθεκτικότητας προκειμένου να μπορούν οι πολίτες στις χώρες που πλήττονται από κρίσεις να ανταποκρίνονται στις κρίσεις αυτές. Χρειαζόμαστε όμως και τον κατάλληλο συντονισμό πριν τη δράση μας και μετά τη δράση μας. Αναφέρθηκα σε τέσσερις κύριους τομείς στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Πρέπει να επικεντρωθούμε τόσο στο πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε άμεσες κρίσεις, αλλά αυτό που πρέπει να μας απασχολεί στη συνέχεια είναι πώς θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τα ωφέλη της ανθρωπιστικής βοήθειας που δίνουμε βραχυπρόθεσμα, δηλαδή η ανθρωπιστική βοήθεια να μεταλλαχθεί στη συνέχεια σε αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις πολύ πλήρες, πλήρης οι απαντήσεις. Έχουμε πολύ δουλειά στο σε εξάμεινο. Η Προεδρία σας ξέρουμε ότι έχει αποφασιστικά εμπλακεί σε όλες τις εκκρεμίε διαδικασίες. Με πολύ χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι θα ξαναρχίσουμε στις 3 με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα μας μιλήσει για το πώς συμβάλλει η ΕΤΕ στην ανθρωπιστική, στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια, συμπληρωματικό δηλαδή των όσων ακούσαμε το πρωί και από τον Όσα. Να είστε εδώ παρόντες και βέβαια μην ξεχάσετε στις 5.30 τις ψηφοφορίες. 12.30 έχουμε τους συντονιστές με γεύμα στο, στην αίθουσα υπαριθμών 2. Η λυπή, καλή σας όρεξη.